Συνάδελφοι, αρχίζουμε τη συνεδρίαση. Θα κάνουμε κάποιες ηλεκτρονικές ψηφορίες στην αρχή. Ας κάνουμε πρώτα-πρώτα ένα τεστ για τις συσκευές ηλεκτρονικής ψηφορίας. Ψηφίστε ό,τι σας έρχεται. Has, has everybody voted? Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίες. Α, δεν λειτουργεί η συσκευή σας. Ας ξαναδοκιμάσουμε. Ψηφίστε πάλι. Για δοκιμή. We are missing some members, but uh, I guess they are coming. Mm. Two more. One more. Λείπουν βέβαια κάποιοι συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος λείπει. Πέρας ψηφοφορίας. Στη μέση διάταξη πρώτα-πρώτα προβλέπεται το σημείο 9 έκθεση Norbert Neuser. Θέλω να μας πει δύο λόγια πριν ψηφίσουμε. Όχι, ευχαριστώ. Οπότε να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Δεν έχουμε τροπολογίες. Μόνο μία ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Ονομαστική είναι. Α, είναι ονομαστική. On Δεν προβλέπεται παρατήρηση στην λίστα της ψηφοφορίας. Τίποτε ονομαστική. Καλά ονομαστική. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκανία πέρα, ένας κατά, καμία εποχή. Εγκρίνεται η έκθεση. The second one uh, is also a report by... Δεύτερη ψηφοφορία και αυτό το κείμενο του Norbert ε, Νόιζερ σχέδιο εκθέσεως και αρχίζουμε την ψηφοφορία. 25 τροπολογίες. Θα ψηφιστούν μία προς μία. Επτά. Διανατάσεις της χειρός. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Ε, ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 16 Ζητείτε ηλεκτρονικός έλεγχος για το 15. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Και εγκρίνεται. Άρα ήταν καλή ιδέα να κάνουμε τον έλεγχο 16 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 10 17. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Θα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Τώρα ψηφίζουμε. Να δούμε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Όχι, όχι, εγκρίνεται λέει ο πρώτος. Συγγνώμη. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψήφισμα. Πέρας. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. 24 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στη συνέχεια έχουμε τις ψηφορίες για τις ειδωλικές παραγράφους. Πρώτη τροπολογία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η επομένη. Έκθεση Μακάβων. Η εφαρμογή των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Έχουν αποσυρθεί κάποιες τροπολογίες. Ας αρχίσουμε την ψηφοφορία. Τροπολογίες 12 και 13 έχουν αποσυρθεί 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 έχει αποσυρθεί. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 καταπίπτει. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 40 καταπίπτει. Πάμε τότε στην 19 υπέρ. Κατά. Αποχές να την ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Έναρξη ψηφοφορίας. Δεν δουλεύει ένα μηχάνημα. Έχω, πρόβλημα με τη συσκευή μου. Πάντως ψηφίζω όχι. Πέρα ψηφοφορίας. καταψήφισε. Συνεπώς απορρίπτεται η συγκεκριμένη τροπολογία. Μήπως μπορείτε να μετακινηθείτε σε άλλη θέση. Ναι, ναι, το έκανα μόλις. Τροπολογία 20, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος επίσης. Έναξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Είδατε, κάθε ψήφος μετράει εδώ. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ηλεκτρονικός της 24. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 είχε αποσυρθεί. Τροπολογία 27 πρέπει να την ψηφίσουμε γιατί 25 κα, καταψηφίστηκε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά έλεγχος έναρξη ψηφοφορίας ψηφίσατε όλοι πέρας Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 και 34 έχουν αποσυρθεί. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τις αιτιολογικές σκέψεις τώρα. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε τροπολογίες έχουν αποσυρθεί. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα ηλεκτρονικός το σύνολο του κειμένου. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρα. is Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα σε ένα σχέδιο προφορικής ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Έναρξη. Πέρας. Γκρίνεται. Συνεχίζουμε. Έκθεση του κυρίου Φρουντζούλιτσα. Νομοδότηση για την ετήσια έκθεση εφαρμογής της κοινή εμπορικής πολιτικής. Θέλετε να πάρετε το λόγο ως εισηγητής, κύριε Φουντζούλητσα. Όχι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, συμβαστική 1, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία... τέσσερα πέφτουν, ε, καταπίπτουν όλες μέχρι την 8. 8 λοιπόν, υπέρ, κατά. <coughs> συγγνώμη, συγγνώμη, ξέχασα τη συμβιβαστική 2, λέει ο πρόεδρος. Υπέρ, κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ε, κάποιος δεν έχει ψηφίσει. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. What is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στη συμβιβαστική 2α. Vote is... Ah. Yeah. The is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 9. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος, εντάξει. What is closed. Πέρας. Πέρας. Εντάξει, ψηφίστε όλοι. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Uh, Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκατρία, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 13. Close the vote. Πέρας. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. It was carried. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 15. Τις 15. Κάποιος δεν ψηφίζει. One Κάποιος δεν ψηφίζει. Δύο δεν έχουν ψηφίσει. Πρέπει όμως να κλείσω την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. So you want to take it again. Θέλετε να ξαναψηφίσουμε δηλαδή. Okay. Let's be generous and vote. Ας είμαστε γενναιόδοροι, να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Κύριε Πρόεδρε. Μου φαίνεται ότι εγκρίναμε τη συμβιβαστική τρία. Όχι. Α, απορρίφθηκε. Α, τότε καλά. Λοιπόν, άρα Πού είμαστε τώρα, στη 16? Ναι, ναι, να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στη 16. Πέρας. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Σας παρακαλώ, σηκώνετε τα χέρια. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18. Α, να ελέγξουμε τη 17. Εντάξει. Πέρας. Απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές Έλεγχος. Έλεγχος στις 19. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος της συμβιβαστικής 4. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος της 23. Closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έρεγχος. Δύσκολη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν, καταπίπτουν τρεις τροπολογίες και πάμε στην 28. Υπέρ. Α, δύο τμήματα, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Έλεγχος, έλεγχος. Το πρώτο του πρώτου τμήματος 28. Πέρας. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Α, έλεγχος. Έλεγχος του δεύτερου τμήματος της 28. Πέρας της ψηφοφορία Απορρίπτεται. 29. Α, όχι, όχι, λέει ο πρόεδρος, συγγνώμη, ε, του συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Στη συμβιβαστική 7 πάμε. Ναι, ευχαριστώ πολύ που με βοηθάτε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. Άρα πηγαίνουμε στην 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές έλεγχος τη 46 Έναρξη ψηφοφορίας. Ακόμα παραμένει ανοιχτή η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Και πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία, στο σύνολο του ψηφίσματος, όπως έχει τροποποιηθεί, η ηλεκτρονική ψηφοφορία έναρξη. The vote is uh, closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Σιγητά. Πάμε τώρα, αφού τελειώσαμε την ψηφοφορία, συνεχίζουμε. Έχουμε στην ημερήσια διάταξη το σημείο 14 την παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών συμπεριλαμβανομένης αρπαγής γης. Colleagues. We now have come to the exchange of views on our draft opinion on the violation. τα δικαιώματα των ε, γενών ε, και το θέμα της αρπαγής γης, ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για την ε, Επιτροπή μας. Βεβαίως δεν είμαστε η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπής, και η ψηφοφορία θα γίνει στις 23 και 24 Απριλίου. Η Μαρία Χόιμπο είναι αρμόδια για την ε, γνωμοδότησή μας. Σου δίνω το λόγο για να την παρουσιάσεις. Σας παρακαλώ πολύ εγκαταλείψετε την αίθουσα με ησυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω ως εξή Στις 17 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κένια υποχρεώθηκε να σταματήσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Γιατί αυτό που μάθαμε τότε είναι ότι υπήρχαν βία επεισόδια και δολοφονίες και σύμφωνα με τις ε, υπηρεσίες ε, της Κένιας μάθαμε ότι υπήρχε βίαιη επίθεση κατά Ιθαγενών στην Κένια με σκοπό να ελευθερωθούν στη δυτική περιοχή της Κένιας, εκεί δηλαδή που υπήρχε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα της Κένιας, μια ολόκληρη περιοχή με αποτέλεσμα να υπάρξουν ε, τραυματίες ε, και ένας νεκρός. Ήταν ε, ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ήδη ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο και οι ΜΚΟ που συμμετείχαν λένε ότι ακριβώς ε, αυτό που συνέβη είναι ότι μετά το ξεκίνημα αυτού του προγράμματος άρχισε οι, άρχισαν οι διώξεις και τα βία επεισόδια κατά των πληθυσμών. Γνωρίζω αρκετές ε, λεπτομέρειες για το τι συνέβη, αλλά θα ήθελα να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Αυτό είναι ένα μεταξύ άλλων παραδειγμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, όπως ξέρετε, αφορά και άλλες περιοχές και άλλους λαούς και πολλές φορές παραβιάζονται τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό να σεβαστούμε το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων στην γη τους στη, ιδιαίτερα στις περιοχές που ζουν εδώ και αιώνες. Το θέμα λοιπόν της γης είναι πάρα πολύ σημαντικό και της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων πρόσβασης. Βλέπουμε ότι πολλές φορές αυτοί οι λαοί βρίσκονται εκεί και ζουν στην περιοχή αυτή, όχι μόνο στην Κένια, αλλά σε πολλές ε, περιοχές ε, του κόσμου, ανήκουν σε αυτή τη γη αιώνες, χρόνια, πολύ πιο παλιά, δηλαδή η δική τους παρουσία είναι πολύ αρχαιότερη από αυτή των σημερινών ιδιοκτητών. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι που θέλουν να αγοράσουν ή έχουν αγοράσει ή θέλουν να εκμεταλλευτούν τις περιοχές αυτές είναι επιχειρήσεις ή ιδιοκτήτες ε, πολυεθνικές που πραγματικά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η φυσική πόρη αυτών των περιοχών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια προστασία νομική, προετοιμασμένη, που να λαμβάνει η χώρα μετά από την ε, ενημέρωση των ε, κατοίκων, μετά από την ε, σωστή ενημέρωση και την συμμετοχή και των ε, κατοίκων της περιοχής. Όλες λοιπόν οι νομικές ρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και ε, τις επιθυμίες και την προστασία των τοπικών πληθυσμών. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι το παράδειγμα της Κένιας δεν είναι μοναδικό, δεν είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει συμβεί πουθενά αλλού. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πώς θα προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει πιο απαιτητικούς κανόνες. Όσον αφορά τώρα τις επενδύσεις, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρουμε ότι το θέμα των ε, επενδύσεων στο εξωτερικό με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πριν από μερικούς μήνες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όλοι οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την ύπαρξη τέτοιων πληθυσμών, τα δικαιώματά τους και βεβαίως στην έκθεσή μου, θέλω, στην γνωμοδότησή μου θέλω να συμπεριλάβω και αυτές τις ε, διατάξεις, τις διευθετήσεις τις οποίες έχουμε ήδη λάβει υπόψη μας. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα δικαιώματα των πληθυσμών αυτών. Πρόκειται για ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο και με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες ζωής, στη φτώχεια. Θα ήθελα λοιπόν να συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις πτυχές του προβλήματος στο κείμενο που θα υποβάλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον ε, παρατηρήσεις και σχόλια. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Ο κύριος Βίλαντ είναι ο πρώτος σκιώδης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, γιατί συμφωνώ απολύτως με τη συνάδελφο. Την ευχαριστώ καταρχήν για την εξαιρετική της εργασία και τον συνάδελφο που είναι ο κύριος εισηγητής. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις, κυρίως γλωσσικές θέματα διατύπωσης. Νομίζω ότι συμφωνούμε καταρχήν και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε λίγες και αρκετά συνενετικές συμβιβαστικές προτάσεις. Νομίζω ότι το νομικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που έχει απασχολήσει και τα Ηνωμένα Έθνη και νομίζω ότι πραγματικά οι επιχειρήσεις θα πρέπει εδώ να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε φορά που υπάρχουν ε, τοπικοί πληθυσμοί δεν μπορούν να αγνοούν την ύπαρξή τους και τις ε, ε, ιδιαιτερότητες τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι η Μαρία Νόχελ. Μα όχι, η Λόλα Σάντσες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Καμπών στη Γουατεμάλα μια ηθογενής είναι φυλακισμένη γιατί κατήγγειλε τόσο γίνονται εκεί για κάποια μέτρα ε, καταστολής για το ότι έχουν αποστραγγίσει το ποτάμι και φτύχονται χιλιάδες. Πάει όλο το ποτάμι και έχουμε την κόμπρα η οποία είναι της Αφέση, μια θηγατρική που είναι ε, ιδιοκτησία του Φλωρεντίνου Πέρεθ του του Ισπανού και έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια ε, για να πάρουν ε, βιοκαύσιμα και πάρα πολλοί έχουν φύγει από αυτό χιλιάδες και έχουμε δεκάδες από γεωτρήσεις ε, έχουμε ε, κολόνες για τον ηλεκτρισμό, αυτοκινητόδρομους, το περιβάλλον και όλα αυτά τα κάνει η Repsol και η BBVA, η Ισπανική Τράπεζα. Στην Ονδούρας η Κάθερες έχει φυλακιστεί και μετά ε, ε, ε, δολοφονήθηκε γιατί ήθελε να αγωνιστεί κατά κάποιων έργων Ολλανδικής Τράπεζας. Και υπάρχει επίσης και ένα φαν φιλανδικό το οποίο υποτίθεται ότι βοηθάει την ανάπτυξη. Αυτά είναι ενδεικτικά παραδείγματα και δεν αφορούν μόνο την αρπαγή γεών και φυσικών πόρων αλλά έτσι αποστρούν τον κόσμο από το ίδιο το νερό που είναι απαραίτητο για την ε, ζωή. Και όποιος διαμαρτύρεται και απαιτεί δικαιοσύνη, δολοφονείται, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί. Έχουμε το 169, το ψήφισμα του, του Γραφείου Εργασίας, αλλά αυτό δεν φτάνει. Θα πρέπει να υπάρξουν επίσημες διαβουλεύσεις πριν ε, οτιδήποτε άλλο εγκριθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιες ε, ρήτης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κεφάλαια για την βιώσιμη ανάπτυξη και λέει ότι αν έχουμε καταπάτηση σύμφωνα με την συμφωνία ε, για καταπάτηση δικαιωμάτων τότε η συμφωνία ε, αναστέλλεται στην ισχύ της. Όμως τελικά αυτά δεν είναι δεσμευτικά. Αυτά είναι μόνο λόγια για να καθισκάσουμε την συνείδησή μας τις προάλλες και ενώ εμείς εδώ τα συζητούσαμε είχαμε χιλιάδες που εθίγησαν κατοντάδες χωριά εθίγησαν στο όνομα μιας στρεβλής ανάπτυξης είχαμε κάποια φρικτά εγκλήματα και οι ηθικοί αυτουργοί κυκλοφορούν με σωματοφύλακες ελεύθεροι άρα θα πρέπει να δούμε πώς η Ένωση θα αποφύγει και τους πολέμους αλλά και πώς θα προωθήσει ανθρώπινα δικαιώματα και γιατί και αυτά είναι συγκρούσεις και αυτά είναι κατάσταση ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι αξίες που θα έπρεπε για την εξωτερική μας εμπορική πολιτική να είναι δεσμευτικές και όχι νεκρό γράμμα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει ένα τέρμα σε αυτά τα εγκλήματα, γιατί είμαστε και εμείς ηθικοί αυτούργοι αυτών. Να προβλέπεται μέσω του ΟΗΕ διεθνής μηχανισμός, μια δεσμευτική ε, συμφωνία να προστατεύει αυτόν τον ε, κόσμο για όλα αυτά τα οποία δικαιούται. Και είμαστε πάρα πολύ ασύνεπείς ότι δεν είναι δεσμευτικές οι λόγω ρήτρες δικαιωμάτων. Έχουμε στρεβλώσει, έχουμε ξεχάσει ε, τις βασικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι τελικά θα βρούμε το σωστό δρόμο. Είμαι αισιόδοξη και επίσης νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε business και εμπόριο χωρίς να καταστρέφουμε τον κόσμο, χωρίς να καταστρέφουμε την ζωή τους. Χρειάζεται όμως πολιτική βούληση για να σταματήσουν αυτές οι κακές πρακτικές, να φρενάρουμε αυτούς τους εγκληματίες επιχειρηματίες και τους κυβερνώντες που επίσης έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα. Η, κυρία Χόιμπουχ έχει την πλήρη υποστήριξή μας. Okay. <coughs> Thank you, Lola. We have one... Ευχαριστώ, Λόλα. Έναν ακόμη σκιώδη εισηγητή έχουμε. Ε, να πόρτα πάρτε το λόγο, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγητής για την ε, έκθεση αυτή. Και επίση έχουμε συναρμοδιότητα. Ε, ο Σύνδεφος Ασής στην ΑΦΕΤ είναι πολύ σημαντικό το θέμα ακριβώς όπως τα είπε και η Λόλα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν κάνει τίποτα τώρα γιατί δεν κάνει τίποτα για να σταματήσουν ε, αυτά τα παράνομα ε, στα οποία προβαίνουν οι πολυεθνικές. Άρα θα πρέπει να έχουμε πολιτικές, διεθνή συνεργασία και κάτι να κάνουμε και για τους ανηλίκους που πάσχουν από κάποια αναπηρία. Και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δεσμευτική συμφωνία για αυτούς. Να υπάρξουν εγγυήσεις για να αποφύγουμε αυτού του είδους την ε, αρπαγή των λιών, αλλά και να προστατεύσουμε τους ε, ανάπηρους που σας προανέφερα. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για όλα αυτά τα οποία γίνονται, για ε, κάποιες εταιρείες εξορυκτικές, για κάποια έργα ανάπτυξης δήθεν, γιατί υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και θα το πράξουμε σε άλλη περίσταση. Κάτε με αυτή η έκθεση είναι σωστή αφετηρία. Να αναλυφθούν οι ενέργειες που πρέπει να προστατεύσουμε τους ηθαγενείς, να προστατευθούν οι φυσικοί πόροι που απειλούνται. Δεν έγινε τίποτα με διμερείς ε, συμφωνίες επενδυτικές. Και το πιο σημαντικό είναι το ότι θα πρέπει να λάβει δεσμευτικά μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις ε, εταιρείε. Χρειάζονται επίσης και κάποιοι μηχανισμοί που να επιβάλλουν κυρώσεις όπου πρέπει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει κάτι σαν μητρό για να δούμε, τη, να καταγράψουμε την δράση των ευρωπαϊκών εταιριών και των πολυεθνικών. Θα πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα των ιθαγενών. Θα πρέπει ό,τι γίνεται να γίνεται με την συνένεσή τους γενικά ό,τι κάνουμε σε τρίτες χώρες. Αυτό όμως να γίνει με νομοθεσία. Οι Ευρωπαίοι είμαστε συνυπεύθυνοι για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των Ιθαγενών. Thank you, Ignacio. Ευχαριστώ, Ιγνάσιο. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Δεν σας γνωρίζω. Δεν σας θυμάμαι μάλλον. Καλημέρα. Λέγομαι Μαρία Νόχελ. Δυστυχώς άργησα γιατί ήμουν σε μια άλλη ε, ψηφοφορία. Θα ήθελα, επειδή είμαι σκιώδης εισηγήτρια, να αναφέρω ένα σημείο που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το θέμα της ευθύνης που έχουμε στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, στον τρόπο που καταναλώνουμε, στον τρόπο που εξάγουμε και στον τρόπο που επενδύουμε. Η δική μας συμπεριφορά εννοείται ότι επηρεάζει μαζί με τους μεγάλους βεβαίως επενδυτές όσον αφορά τις επιπτώσεις για όλους αυτούς τους λαούς οι οποίοι σήμερα βρίσκονται παραπερισμένοι και θύματα αυτής της αρπαγής γης. Και βεβαίως αυτό το λέω γιατί αφορά όλους τους τομείς. Αφορά το θέμα των φυσικών πόρων σε όλους τους τομείς. Και για τα λιεύματα και για τα ορυκτά και για τα δάση και όπως είπαν φαντάζομαι και οι προηγούμενοι ομιλητές η δική μας ευθύνη, η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που αφορούν τις εξαγωγές, σε θέματα που αφορούν τη γενικότερη οικονομική μας πολιτική, την αλληλεία, την δασοκομεία και την ε, πολιτική μας στον τομέα των ε, εξορρυκτικών βιομηχανιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, είστε σκιώδη συγγήτρια για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Θέλει κανένας άλλος συνάδελφος να πάρει το λόγο? Είναι εδώ κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την ΕΕΔ που θα ήθελε να πάρει το λόγο? Please introduce yourself. Παρακαλώ συστηθείτε. Ευχαριστώ. Του Εγκέντ λέγομαι και είμαι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης ε, από το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχαμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε αυτό το σημαντικό σχέδιο έκθεσης, οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Απλώς θα ήθελα να πω ε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ενισχύσει την ε, υποστήριξη των ε, ανθρώπων, των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στο πλαίσιο του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής και θα ήθελα να σας επιστήσω και την προσοχή στο, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου του 2017 τα οποία Επίσης θέτουν τις απειλές και τις παραβιάσεις κατά των αυτοχθόνων πληθυσμών σε σχέση με τα δικαιώματα επί της γης τους, ε, σε προτεραιότητα ε, και τα θεωρεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με την άνηση μεταχείριση που λαμβάνουν οι άνθρωποι αυτοί επειδή έχουμε μία προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα στην αναπτυξιακή συνεργασία και θα έπρεπε αυτό να παραμένει το, ο βασικός φορέας υποστήριξης των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών ε, με, κατά την εφαρμογή του, του προγράμματός μας μέχρι το 2030 θα έπρεπε να ενισχύσουμε ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρίες, ε, του νέους και τα παιδιά. Επίσης, όσοι βρίσκονται σε, σε υποχρεωτικό εκτοπισμό ε, και σε περιοχές συγκρούσεων ε, όσον αφορά την πρόληψη συγκρούσεων και τις ειρηνευτικές διαδικασίες όλα αυτά επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη επίσης τα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπενθυμίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και τις επιχειρήσεις και το αναφέρει σε σχέση με τους αυτόχθονες αυτούς πληθυσμούς. Επίσης αναφερθήκατε σε αυτή τη σημαντική αρχή της πρώτερης συγκατάθεσης. Το Συμβούλιο επανεπισημένει την ε, ε, υποστήριξε της αρχής αυτής λέγοντας ότι ο διάλογος και η διαβούλευση με, ε, τις, ε, με τους πληθυσμούς αυτούς ε, συνεχίζεται σε όλα τα στάδια της εφαρμογής των προγραμμάτων για να εξασφαλιστεί η πλήρη συμμετοχή, του, η συμμετοχή τους και η συγκατάθεσή τους κατά πλήρη και συστηματικό τρόπο. Ήδη από το 2000 13 έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη νομοθεσία που θεωρούν ότι πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που σημαίνει επίσης ότι επηρεάζεται και η εμπορική μας πολιτική και κάθε φορά που έχουμε αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο αυτό, ε, αναφερόμαστε και στα δικαιώματα των ε, αυτοχθόνων πληθυσμών. Αναμένουμε εναγωνίω ε, την κλήρωση τη έκθεσης αυτή, όπως και την περαιτέρω συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Είναι εδώ κανένας από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Όχι. Εντάξει. Είναι κάποιο εδώ. Α, παρακαλώ. Συστηθείτε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Σιλβί Πουλβέρ. Δουλεύω στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ στο Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είμαι υπεύθυνη για το θέμα αυτό των δικαιωμάτων αυτοχθόνων πληθυσμών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές που πήραν το λόγο για να παρουσιάσουν την κατάσταση, την οποία δυστυχώς τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, ειδικότερα στο δικό μας το τμήμα, γιατί διαχειριζόμαστε το μηχανισμό υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε όλο και περισσότερο είναι ότι οι υπερασπιστές αυτοί δολοφονούνται, ε, ειδικότερα εκείνοι που υπερασπίζονται τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, την διατήρηση της γης, ε, και ε, βεβαίως ε, όσοι υπερασπίζονται κυρίως τους αυτόχθονες πληθυσμούς που βρίσκονται σε περιοχές ε, όπου υπάρχουν μεγάλα προβλήματα φυσικών πόρων. Πέντε εκατομμύρια της δημοσιονομικής γραμμής της πρικοδοτημένης για το συγκεκριμένο θέμα έχουν εγκριθεί ε, περιμένουμε να ολοκληρωθεί το, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προγραμμάτων, ε, οι, οι πολιτικές ε, επενδύσεων, τα, οι επιχειρήσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Γενική Διεύθυνση η Άγκρη, όλα αυτά αναφέρθηκαν. Είναι μια τεράστια πρόκληση για μας για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να υπάρξει συνεργασία εσωτερική και εξωτερική. Το καλύτερο παράδειγμα της συνεργασίας αυτής από τότε που εγώ εργάζομαι στην ανάπτυξη είναι το VPA, ε, το οποίο ε, σημαίνει ένα, υπάρχει, ε, περιλαμβάνει ένα εσωτερικό κανονισμό εισαγωγής ξυλίας, κάτι το οποίο δείχνει την συνεργασία εσωτερική και εξωτερική, αυτό που θα ήθελα να πω ολοκληρώνοντας είναι ότι έχουμε αυτή την προσέγγιση τη βασισμένη στα δικαιώματα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε. Ε, είναι πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε στην ε, υλοποίηση των προγραμμάτων επικαθημερινής βάσεως γιατί υπάρχουν τέτοια προγράμματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κίνδυνο για την κοινότητα Σύγκουε στην Κένια, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, ε, ένα πρόγραμμα ε, για το περιβάλλον. Ε, η αντιπροσωπεία νέστηλε κάθε χρηματοδότηση λόγω της τελευταίας δολοφονίας που έγινε τον Ιανουάριο μόνο αυτό έχουμε ως μέσο αντίδρασης. Ε, δεν έχω δει, τουλάχιστον στο δικό μου επίπεδο πληροφόρησης, τόσα χρόνια που δουλεύω στη Γενική Διεύθυνση, δεν έχω βρει μηχανισμό ε, καταγγελίας, ας πούμε, ε, εναντίον μιας ευρωπαϊκής επένδυσης ε, ή ενός προγράμματος αναπτυξιακού, ούτε έχουμε κάποιο μηχανισμό ε, αντιστάθμισης, αποζημίωσης, αποκατάστασης εγώ διάβασα την έκθεση, τη βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, είναι πολύ εξισορροπημένη. Θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ ε, τους ε, συντάκτες της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε μήπως ε, να πείτε κάτι για να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ γιατί δώσατε πολλά παραδείγματα. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι και η έκθεση αυτή αλλά και η γνωμοδότησή μας βασίζεται σε πραγματικά και πολλά τέτοια παραδείγματα. Χαίρομαι που η Επιτροπή διαπιστώνει από μόνη της ότι σήμερα δεν υπάρχει μηχανισμός για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις περιπτώσεις, τις προσφυγές και να αντιδράσουμε. Υπάρχουν άτομα που έχουν πληγεί, είτε πρόκειται για αυτόχθονες πληθυσμούς, είτε πρόκειται για ομάδες ανδρών, γυναικών και παιδιών που πλήττονται από τη δράση μας, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και ακούσαμε πόσο πολλά παραδείγματα υπάρχουν, ότι θα πρέπει να υπάρχουν τρόποι αντίδρασης και ελπίζω ότι δεν θα παραμείνει το θέμα αυτό στο χαρτί σε μια έκθεση, αλλά ότι κάτι θα ακολουθήσει, όπως παραδείγματο χάρη ένας μηχανισμός για να λαμβάνονται υπόψη οι προσφυγές και με έναν αποτελεσματικό τρόπο να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Και νομικά αλλά και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα λάβω υπόψη σας όλες τις παρατηρήσεις. Κύριε Βίλαντ, μιλήσατε για μεγάλη συνένεση για συμβιβασμό. Ελπίζω ότι οι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν θα μπορέσουν να υποστηριχτούν ε, από όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος Μαρία. Ευχαριστώ όλους για τις συνεισφορές σας. Την Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα, στις 5 το απόγευμα είναι η προθεσμία για την υποβολή των ε, τροπολογιών και στις 20 Μαρτίου θα ψηφίσουμε. Ολοκληρώθηκε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο, στο 15, που είναι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Δημοκρατία του Κονγκό. Ο διευθυντής ε, υπεύθυνο για την Αφρική, την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Εντουάρδο Καμινάρα, θα μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. So, I'm going to make a... Οπότε, λέει ο πρόεδρος, θα κάνω εγώ μια σύντομη εισαγωγή, ενώ κάθεται η κυρία Καμιναρά. Είμαστε στο επόμενο σύνδεσμο ε, της ε, ε, Διατάξεως. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη λακή Δημοκρατία του Κονγκό κατάσταση είναι πάρα πολύ ενισχυτική εδώ και πολλά χρόνια και στο Σοβείο Πόλεμο με εκατομμύρια νεκρούς στην Ανατολική χώρα και το 2017 θεωρείται ένα από τα πιο βία χρόνια στην πρόσφατη ιστορία. Και εν μέρει αυτό γιατί η κατάσταση πολιτική είναι ασταθής, έχουμε αύξηση της ε, βίας, ιδίως ε, στο βόρειο και νότιο Κιβού, αλλά και στην επαρχία της Ταγκανίκα και στο Κασάι. Ως αποτέλεσμα, στη χώρα έχουμε ένα σύνολο 4,3 εκατομμυρίων εσωτερικά εκτοπισμένων. Το 2018 είχαμε το πρόγραμμα ανθρωπιστικής ε, αντίδρασης ε, για τη χώρα, οπότε και εκταμιεύτηκαν 1,7 δις δολάρια για να βοηθηθούν 13 εκατομμύρια που είχαν ε, ανάγκη. Η ε, θεώρησε ότι υπάρχει κατάσταση ανάγκης στο επίπεδο 3 και ε, επομένως χρειάζεται η αντίδραση ε, η πιο πλήρης. Αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 2013, παρ' όλα αυτά όμως είμαστε ακόμα σε πάρα πολύ χαμηλή χρηματοδότηση με παγκόσμια κριτήρια. Οπότε φτύσαμε δώσουμε το λόγο στην κυρία Καμινάρα για να μας τα εξηγήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ λοιπόν, που μου δίνετε την ευκαιρία για να τα συζητήσουμε όσον αφορά το Κονγκό. Αυτό που θέλω σήμερα να σας πω αφορούν τρία διαφορετικά σημεία. Πρώτα-πρώτα αυτά τα οποία είδα στην πρόσφατη εκεί επίσκεψή μου για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, κατά δεύτερό λόγο, πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τη δική μας αντίδραση και να σας ενημερώσω για κάποια διάσκεψη που θα οργανώσει για τη χώρα ο ΟΗΕ. Οπότε, η ανθρωπιστική κατάσταση. Να σας διαβάσω τι είπε ο διευθυντής μίας ΜΚΟ σε σχέση με αυτή την ενίσχυση για τη χώρα. Το 2017 ήταν πάρα πολύ άσχημη χρονιά, το 2018 θα είναι χειρότερο. Και από όσα επιτόπου διαπίστωσα, και εγώ θα προσυπέγραφα αυτό το οποίο είπε ο Διευθυντής. Ήδη ακούσατε κάποια στοιχεία. Να σας τα αναλύσω ακόμη περισσότερο. Έχουμε 13 εκατομμύρια που χρειάζονται βοήθεια 7,7 δεν έχουν αρκετή τροφή, σχεδόν 2 εκατομμύρια ανήλικοι έχουν πληγεί από κακή διατροφή και πάνω από 4 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί στο ιστορικό της χώρας ε, που είναι ρεκόρ για την Αφρική και να μην ξεχνούμε ότι περίπου μισό εκατομμύριο ε, Κογκολέζοι βρίσκονται στις ε, γείτονιές χώρες στο Σουδάν, στο Μπορούντι και στις άλλες. Α, και στη Ρουάντα και αλλού. Και ο κόσμος φεύγει και πάει σε χώρες σαν το Νότιο Σουδάν. Ε, μπορείτε να καταλάβετε τότε πόσο απελπισμένη είναι και πόσο μεγάλη είναι η ανθρωπιστική κρίση που είναι σοβαρή και σε εκείνες τις χώρες. Έχουμε διάφορες επιδημίες, ε, έχουμε περιστατικά χολέρας στην Κινσάσα και είχαμε επίσης 55.000 περιστατικά χολέρα στα τέλη του 2017. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να βοηθήσει και να αντιμετωπίσει την χολέρα. Χθε αναφέρθηκε ότι τώρα Κογκολέζοι φεύγουν προς την Ουγγάντα Οπότε πάει και η χολέρα εκεί. Πάνε γιατί έχουν προβλήματα σε Ογκάντα και σε άλλες χώρες, οπότε υπάρχουν και εκεί προβλήματα. Επίσης χρειάζεται προστασία επιγόντως και έχουμε τουλάχιστον 120 ενοπλές ομάδες που δρούν ή στην χώρα. Και αυτό είναι πρόβλημα, όχι μόνο γιατί έχουμε Συγκρούσει στη χώρα, αλλά γιατί έτσι δυσκολεύει και το έργο των ανθρωπιστικών φορέων, γιατί δεν πρέπει να ξέρουμε ποιο κάθε φορά ελέγχει την περιοχή που θέλουμε να έχουμε πρόσβαση. Είναι όλες αυτές οι ομάδε, ομάδε, ε, μεταβάλλεται συνεχεία κατάσταση που το ανθρωπιστικό έργο καθίσταται πολύ δύσκολο και να μην ξεχνούμε. Βέβαια, το πολύ γνωστό θέμα, το μέγεθος του Κονγκό είναι όσο μεγάλο η Δυτική Ευρώπη και είναι και οι γειτονικέ χώρες και επίσης το ότι το Κονγκό αποσταθεροποιεί μεγάλο τμήμα της Υπήρου. Τώρα, αναλάβουμε το πόσο πίεζε ο να σας περιγράψω τι είδα εκεί. Δεν έχουμε όμως χρόνο, οπότε θα επανέλθω όταν έχουμε ερώτα απαντήσεις. Διάφορες παράγοντες ε, ε, συνάντησα στην Κινσάσα, αλλά και αρκετό χρόνο επισκέφθηκα το Κασάι. Άρα εδώ έχουμε όλα τα στοιχεία μιας ανθρωπιστικής καταστροφής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβληματίζεται βαθιά για το ανθρωπιστικό πρόβλημα και όπως ήδη σας ανέφερα αν φτάσουμε να κάνουμε προγνωστικά για το 18 ε, μάλλον θα καταλήξουμε ότι η κατάσταση δεν θα είναι και πολύ καλύτερη. Δύο λόγια τώρα για το Κασάι. Γιατί εκεί πήγα περισσότερο. Πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι δεν επρόκειτο για ανθρωπιστική κρίση το 2016. Μιλούμε για το τι γινόταν το 2016 στο Βορείο Κιβού. Ναι, εκεί υπήρχε ανθρωπιστική κρίση. Στο Κασάι όμως δεν υπήρχε. Τώρα η ανθρωπιστική κρίση σοβεί και στο Κασάι. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο που φεύγουν από τα σπίτια τους περίπου οι μισοί προσπάθησαν ή να επιστρέψουν ή ήδη επέστρεψαν στο μεταξύ. Αλλά χάθηκε η εισόδια, έχουν καεί σχολεία, σπίτια, νοσοκομεία και επίσης η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες της χώρας σε σχέση με το τι απαιτείται. Κάνει την μπορεί η κοινότητα. Έχουμε όμω συνδυασμό πολιτική κρίση, κρίση υπανάπτυξη, ανθρωπιστική κρίση. Όλα ταυτοχρόνω. Και τα ε, υπόλοιπα στοιχεία ε, συντρέχουν και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τους αδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης για την Ανάπτυξη. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι που διατίθενται θα αξιοποιούν όσο γίνεται περισσότερο. Και ένας από τους τομείς όπου προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε είναι το τομέας της υγείας που καυτό θέμα στο Κονγκό. Πήγα σε ένα νοσοκομείο στο Κασά. Ήταν το μόνο νοσοκομείο που σε 20 200 χιλιόμετρων είχε ένα χειρούργο. Το μόνο, το μόνο νοσοκομείο. Μιλάμε για 200 χιλιόμετρα. Η περισμένη χρηματοδότηση του παρελθόντος προέρχεται από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά πια δεν φτάνει εκεί. Πώς να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο χωρίς να υπάρξει χρηματοδότηση για τη συντήρησή του. Κάτι άλλο τώρα, το οποίο έμαθα στην επίσκεψη και θα πάμε εδώ σε κάτι άλλο, ότι περί τα τέλη του 17 όλες οι ενδείξεις κατέτειναν στο ότι πηγαίναμε προς μείωση των εκτοπισμένων, προς σταθεροποίηση, λιγότερες σύγκρουσεις. Τέλος Ιανουαρίου πήγα. Τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου όμως είχαμε αύξηση των συγκρούσεων, περισσότερους εκτοπισμένους και τα είπαν αυτά όσοι ήταν στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεχόταν όλο και περισσότερους τραυματίες. Um, uh, Οπότε είχαμε την πτώση αλλά κατόπιν είχαμε και την απότομη αύξηση των αρνητικών χαρακτηριστικών. Είχαμε ταχεία αντίδραση. Το Νοέμβριο το Συμβούλιο κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα για τη χώρα. Και είπαμε ότι οπωσδήποτε θα πρέπει ο ΙΕ να αναβαθμίσει τι προσπαθίε του, τον συντονισμό του για να αντιμετωπίσει τη κατάσταση. Και από τότε σημειώθηκε πρόοδο. Τώρα έχουμε κάποιον ειδικό εκπρόσωπο τον Κιμπόλτο πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα. Αυτός ανέλαβε καθηκοντά του τον Ιανουάριο. Οπότε βλέπουμε ότι ο ΟΗΕ αναβάθμισε τις προσπαθίες του. Και, όπως ήδη ακούσατε από τον Πρόεδρο, φτάσαμε σε βαθμό ε, αντίδρασης και αντίστοιχα κρίσης του βαθμού, της βαθμίδας 3. Δηλαδή στο ανώτοτο. του. Όσον αφορά τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Αυτό συνεισφυσχεί για εξάμεινο, 20 Απριλίου λίγη. Η δική ανακοίνωση και αυτό αφορούσε όχι όλη τη χώρα, τρεις. Τον Νότιο Κιβού, την Ταγκανίκα και το Κασάη, εκεί που ήμουν εγώ. Και μην ξεχνούμε και το βόρειο Κιβού, οπότε εκεί πέρα, πέρα είναι κάποιοι δείκτες που ήταν πολύ χειρότεροι. Αλλά μια που αυτό κρατάει εκεί πολλά χρόνια, θεωρήσαμε ότι αυτό ήδη έχει ληφθεί υπόψη από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και σούλεγαν περισσότερο με τις νέες ανθρωπιστικές κρίσεις. Επίσης, Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ θεωρήθηκε ότι έχει πρόβλημα χρηματοδότησης. Και ότι έχει συρρυκνωθεί. Οπότε, στα σημερινά του Συμβουλίου και επιβεβαίως ε, από την εικόνα μου επιτόπου ότι αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για τη χώρα. το Κασάι, ήταν όλα ένα και λιγότεροι. Έτσι και λίγοι ήταν και κάπως βοηθούν ούτως ώστε να συγκρατήσουν κάπως ε, οι συγκρούσεις για να μην ε, ξεφύγουν από κάθε έλεγχο. Υπάρχει και εντολή προστασία προς την ερθική δύναμη. επομένω η κατάσταση στην ε, χώρα αφορά κρίση προστασίας. Τρίτον, Θέλω να σας πω για την ανθρωπιστική διάσκεψη στην χώρα. Έχουν γίνει διάφορες ανταλλαγές, απόψε διάφορες επαφές πριν τα Χριστούγεννα και έχω εμπλακεί και εγώ ούτως ώστε να γνωστοποιηθεί το πώς έχει καταστάσει και τώρα έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δωρητές στις 13 Απριλίου στην Γενέβη πρόκειται να κάνουν αυτή την διάσκεψη. Εκεί θα είναι παρόν ο Επίτροπος ε, Στυλιανίδης και θα με τον Μαρκ Λόκοκ, τον επικεφαλής της ε, Ότσα και με τον Ολλανδό Υπουργό Εξωτερικών, την Υπουργό, την κυρία Συγκριτικά. Ενδεχομένω. θα υπάρχει και τέταρτο συμπρόεδρο. Όλα αυτά ούτω ώστε να προβληθεί περισσότερο αυτή η κρίση και να υπάρξει προσπάθεια για περισσότερους πόρους. Οπότε, ακριβώ το μέτωπο αυτό τη μοντότητα είναι ε, πάρα πολύ μεγάλη και έχουμε διπλασιάσει τη βοήθειά μας. Πάμε τα 2,8 δι. Αλλά είναι μια πιο μεγάλη κρίση σε όλο τον κόσμο. Άρα χρειάζεται η ανθρωπιστική προσπάθεια να είναι παγκόσμια. και θα είναι πρόβλημα ακριβώ επειδή έχουν πολλέ κρίσει να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο βοήθεια. Το 2017 η Ένωση και τα κράτη-μέλη έδωσαν 200 εκατομμύρια δολάρια στο Κονγκό για την κρίση και τότε είχαμε πρόγραμμα 800 εκατομμυρίων. Οπότε όλη μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έδωσε το 25% των όσων έπρεπε να δοθούν. Η Επιτροπή ενήργησε για την χρηματοδότηση και ο Επίτροπος θα επισκεφθεί την χώρα πριν τη διάσκεψη για να μπορεί να έχει προσωπική άποψη για το πώς έχει κατάσταση. Για να μπορέσει ενδεχομένω να ανακοινώσει κάποια συγκεκριμένα ποσά για το τι θα κάνουμε για την κρίση το 18. Εδώ θα βάλω τελεία και βεβαίως περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Και τώρα οι συνάδελφοι μπορούν να πάρουν το λόγο. Μόνιμος εισηγητής μας για την ανθρωπιστική βοήθεια, ο Ενρίκη Γερέλο Σαλόμ, θα λάβει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ όχι μόνο που ήρθατε σήμερα και που μας μιλήσατε, αλλά σας ευχαριστώ και για την συνεχή σας παρουσία στο έργο μας. Να μας μιλήσετε για αυτές τις ανθρωπιστικές τραγωδίες σε σχέση με το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Οπότε και ε, προκειμένου είναι μία από τις πιο μεγάλες κρίσεις που συζητούμε τώρα και νομίζω ότι το σύνολο των συναδέλφων στην Επιτροπή μας σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση και ευχαριστούμε για όλα σας τα ταξίδια επί τόπου για να δείτε στην πράξη όλη αυτή τη δυστυχία, όλες τις ανάγκες που έχουν αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων για το πόσο τους λείπουν τα προς το ζήν. Δηλαδή, μας λέγατε ότι το 18 θα είναι χειρότερο από το 17 και πρόκειται για κριτήριο και πρόκειται για το πού έχουν φτάσει οι ανθρωπικές κρίσεις στον κόσμο. Γιατί όλο ένα και περισσότερο οι κρίσεις δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα, αλλά χρόνιο, μόνιμο. Ε, αυτό είναι ακόμα ένα πρόβλημα από πλευράς πόρων. Ακριβώς όπως μας τα είπατε στο τέλος της σύγκριση ε, σας, ότι αυτά που είχαν προγραμματιστεί ε, αυτά που έχουν προγραμματιστεί για το 2018 ε, είναι πάρα πολλά χρήματα, περίπου 1.800.000 ε, δις. Άρα θα πρέπει να συνδυαστούμε, να δούμε, τέλο πάντων να υπόψη πόσο πρέπει να δώσουμε σε άλλε κρίσεις στον κόσμο. Μα όταν είναι χρόνιες οι κρίσεις, αυτό πάει να πει ότι ένα μεγάλο τμήμα των διαθέσιμων πόρων θα πρέπει να κατευθυνθούν προς υπάρχουσες κρίσεις και η αντίδρασή μας για τις καινούργιες κρίσεις καθίσταται πιο δύσκολη. Μας είπατε τι γίνεται ανά περιφέρεια της χώρας, μας είπατε ότι είναι σε επίπεδο 3, επίπεδο 3 είναι το ανώτατο, το, το, το χειρότερο και έχουμε ένα σωρό κρίσεις σε όλο τον κόσμο που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση σήμερα. Συρία, Σουδάν, Φερρυπίν και θα ήθελα να πω ότι σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές με κρίση τα πράγματα προβάλλονται στην Ευρώπη. Προκαλούν, αγγίζουν την ευαισθησία των Ευρωπαίων γιατί μας αγγίζουν άμεσα μια που για τα σύνορά μα, για τις χώρε χώρες μας ε, έχουν συνέπειε όπω γίνεται με τη Συρία. Ε, Επίση έχουμε τεράστια κρίση στο κέρα Αφρική, έχουμε την κρίση του Κονγκό που αφορούν δεκάδες εκατομμύριων. Όμω είμαστε εμεί μακριά από αυτού, γιατί είναι απομακρυσμένε αυτέ οι κρίσει αυτέ οι περιοχέ γεωγραφικά. Επομένω. έχει σημασία αυτό το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του να είναι παρούσα για επιτόπου να μας ενημερώνει και να αναλαμβάνει τέτοιο πρωταγωνιστικό ρόλο όπως θα κάνει και στην συνάντηση της Γενέβης. Και όπως είπατε, στόχος είναι να αποσπαστούν, να, να, να εξασφαλιστούν πόροι, να προβληθεί η κρίση. Άρα νομίζω ότι σε καλό δρόμο είσαστε. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω κάτι. Μας είπατε δύο λόγια για τη σχέση μεταξύ ανθρωπιστικής ε, βοήθειας και ανάπτυξης. Αν θέλετε πέστε μας δύο λόγια παραπάνω. Επίσης δεύτερον, πέστε μου, εάν η πολιτική συγκυρία στη χώρα, μια που μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα γίνουν κάποιες εκλογές, αν γίνουν θα βοηθήσουν ή θα τα κάνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα όσον αφορά τη βοήθεια την ανθρωπιστική. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε πρώτα όλε τι ερωτήσεις και μετά θα απαντήσετε στο τέλος. Κύριε Ντέβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάντοτε το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, πάντοτε πρωτοστασή και στα 18 χρόνια που εγώ συμμετέχω σε αυτή την Επιτροπή, έχει κάνει πάντοτε πάρα πολύ καλή δουλειά ως προς την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την πρόληψη ε, της, του, του, του να υποφέρει ο κόσμος. Το ζήτημα λοιπόν του Κονγκό έχει πλέον γίνει πολύ σημαντικό πριν από 15 15 χρόνια πρώτη φορά άρχισα να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Ε, προσπαθήσαμε να διώξουμε όλους όσους ε, είχαν, ε, ήταν υπεύθυνοι και μερικοί μάλιστα μερικών υπόθεση έφτασε μέχρι και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το να έχουμε λοιπόν αυτό το ενημερωτικό δελτίο μπροστά μας ε, σημαίνει ότι έχουμε ένα παράδειγμα του τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Συνοψίζει ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα που είναι όμως όχι μια θεομηνία, δεν είναι ένα τσουνάμι, δεν είναι ένας σεισμός, είναι κάτι το οποίο έχει προέλθει από τον άνθρωπο. Συνεπώς η Επιτροπή αυτή και οι φορολογούμενοι μας πρέπει να γνωρίζουν ποιο το ξεκίνησε όλο αυτό, ποιο είναι ο υπεύθυνο, ποιο πρέπει να συλληφθεί και προς πρέπει να δικαστεί γιατί τα χρήματα των φορολογουμένων μας ε, εξακολουθούν να πηγαίνουν σε ζώνες συγκρούσεων των ανθρώπων αυτών οι οποίοι δημιουργούν αυτές τις συγκρούσεις για προσωπικό κέρδος. Ε, όχι επειδή δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, αλλά γιατί σε αυτή την περιοχή, ειδικότερα στην περιοχή του Κιμπού και την περιοχή δίπλα στη Ρουάντα, υπάρχουν τεράστιοι, ε, τερά, τεράστιοι πόροι φυσικοί λοιπόν, ε, και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίξουμε, να υποστηρίζουμε και να βοηθούμε τον κόσμο απλώ και μόνο γιατί βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση όταν η ηγεσία των ανθρώπων αυτών δημιουργεί εκείνη τα προβλήματα για το λαό τη. Ε, πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο επιτόπου ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο και ε, πρέπει να ε, βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς και πρέπει να λογοδοτήσουμε Ρωτείτε σε εμά να μα ενημερώνετε για αυτά που γνωρίζετε, για να μπορούμε και εμεί να ενημερώνουμε τον κόσμο εκεί. Πρόεδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε Σίλκι Έγκε. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την εισήγηση, αλλά στο Κονγκό η κατάσταση είναι τέτοια που την γνωρίζω καλά. Ξέρω λοιπόν όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί και άκουσα την έργα που μας μίλησε προηγουμένως για την κρίση, για τις συγκρούσεις, όλα αυτά τα οποία ανάλογα με την απόσταση έχουν μικρότερη ή μεγαλύτερη ε, επίπτωση σε εμά. Είναι πολλές οι αιτίες της κρίσης στο Κονγκό, είναι η οικονομική κρίση, η πολιτική κρίση, το ένα προκαλεί το άλλο και τελικά καταλήξαμε στην ανθρωπιστική κρίση. Δεν με κάποια κρίση χαμηλής έντασης, γιατί έχουμε όμως τελικά 6 εκατομμύρια, από ό,τι λένε, νεκρούς. Όμως ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα πάμε για τα 10 εκατομμύρια θυμάτων από το 96 μέχρι σήμερα που έχει κρατήσει αυτή η διαδρομή. Πρόκειται για εκατομμύρια νεκρών από ό,τι φαίνεται είναι ένα τέτοιο νούμερο που επιβάλλεται κανείς να παρέμβει. Βέβαια είναι και το θέμα των φυσικών ε, πόρων και η αυτό όπως δεν έχει γίνει τίποτα και αυτό όμως που συμβαίνει στη χώρα είναι παράδειγμα το πώς τα οικονομικά συμφέροντα πολλές φορές σε πολλές ε, χώρες ε, δίνουν το πάνω χέρι στο, στα, στα οικονομικά και όχι στην ανθρώπινη ζωή. Επομένω δεν γίνεται τίποτα παρά τα 10 εκατομμύρια των ε, νεκρών. Ε, όλοι αυτοί οι νεκροί απαιτούν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτή η ανθρωπιστική κρίση είναι ε, κάτι που έφτασε τώρα και στο Κασάι, αλλά ε, εκεί έχουμε το κοβάλτιο που είναι ε, μεταλλό που θα χρησιμοποιηθεί πολύ στο άμεσο μέλλον. Θα φέρει επανάσταση τεχνολογική και προέρχεται από την Κατάγκα. Έχουμε τώρα φυγή πολλών που πηγαίνουν στην Ζάμπια από εκεί και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Είναι πρόσφυγες που έρχονται από το Κονγκό λόγω της ανθρωπικής κρίσης. Και μέχρι πότε θα αντιμετωπίζουμε την κατάσταση σαν ανθρωπιστική κατάσταση ενώ έχει άμεση σχέση με κάποια πολιτική κατάσταση και με ένα καθεστώς που επιβάλλει στον κόσμο να αποδεχθεί την κυβέρνηση αυτή ενώ προξενεί περισσότερο κακό παρακαλώ. Και λόγω αυτών των ε, συμφωνιών του Αγίου Σιλβέστρου έμεινε ο Καμπυλά στην εξουσία. Και μέχρι σήμερα έχουμε τέτοιες ε, συμφωνίες που συνήφθησαν για να δώσουν κάποια λύση ανταυτού όμως είναι αντισταγματικές ε, και τελευταία φορά πήγαμε στη συμφωνία του 16 ε, όμως δεν τηρήθηκαν ε, ε έγινε μια παράταση για τέλος του 17 τώρα πάμε για 18 δεν πρόκειται για συμφωνίες αλλά για φάρσα είπαμε να πανεύουμε για να λυθεί η πολιτική κρίση γιατί αυτή η πολιτική κρίση ωφελεί τελικά όλα τα οικονομικά συμφέροντα και επομένω, νομίζω ότι για δεύτερη φορά δεν κάνουμε τίποτα. Και τώρα μέσω της βοηθείας του ΚΑΣΑΙ θα κάνουμε αυτή τη διάσκεψη των ε, δανειστών. Αλλά σε ποιον θα πάνε τα χρήματα που θα μαζευτούν, θα πάμε σε αυτούς τους διεφθαρμένους. Πώς θα γίνει η διαχείριση, τελικά στον κόσμο καταλήγουν πενταροδεκάρες. Ποιος θα εγγυηθεί για την αξιοποίηση αυτών των χρημάτων τι ρόλο θα έχει το ε, κοινοβούλιο, πώς θα ωφεληθούν, πώς θα πάρουν κάποια χρήματα αυτοί που κρύβονται στη ζούγκλα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανένας άλλος να πάρει το λόγο. Αν όχι, θα ήθελα να ρωτήσω αν η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ θέλει να πάρει το λόγο. Είναι κανείς εδώ που την εκπροσωπεί. Όχι. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Καμινάρα. Με πολύ χαρά θα ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω. Νομίζω ότι κάποιες ερωτήσεις ε, αφορούν ε, στην ευθύνη του κράτους ε, ενώπιον ε, του ντόπιου πληθυσμού και αναφέρθηκα σε αυτό όταν μίλησα για το ζήτημα της ε, ε, έλλειψης ιατροφαρμακευτικής περιθελψής. Κατά την αποστολή στην οποία πήγα εκεί, μπόρεσα από μόνη μου να καταλάβω πόσο δύσκολο είναι να πάει κανείς να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στην δημοκρατία του Κονγκό, ε, πόσο δύσκολο είναι να φορολογήσει κανείς ε, ε, τα πάντα, την προσγείωση, την απογείωση του αεροπλάνου, όπου και να πάει κανείς. Υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και οποιοδήποτε άλλος, πρέπει να περάσει από γραφειοκρατικά εμπόδια κατά την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και σε μια συνάντηση που είχαμε την νέα, κυβέρνηση του Κασάι, ήταν ένα από τα βασικά βασικά ζητήματα τα οποία έθεσα. Δηλαδή, οι υπεύθυνοι ανθρωπιστικής βοήθειας είναι εκεί για να βοηθήσουν τον κόσμο. Ε, προσπαθήστε να μας βοηθήσετε να το κάνουμε και εμείς με λιγότερο δαπανηρό και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κύριος Δέβα, εκτός μικροφώνου δυστυχώς. Δεν λέω ότι βγάζουν λεφτά από αυτό είναι η απάντηση. Ε, το ζήτημα είναι ότι είναι έτσι η κατάσταση ώστε για να μπορέσει κανείς να έχει πρόσβαση ε, στο αεροδρόμιο ε, κάποιος ε, πρέπει να πληρώσει κάτι και φυσικά η ανθρωπιστική βοήθεια δεν εξαιρείται από αυτό. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για την ανθρωπιστική κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να ε, υπερβούμε όλα αυτά τα ε, ζητήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τα ζητήματα ασφαλείας επίσης, γιατί η χώρα αυτή είναι μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές. Ε, εχθές ή προχθές υπήρξε μάλιστα και αναφορά μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που δούλευε στην περιοχή των Κιβού ε, και μάλιστα ε, κάποιος από την αποστολή απήχθη και ε, δολοφονήθηκε. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολη η κατάσταση επιτόπου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκτήσει κανείς πρόσβαση και να εξασφαλίσει κανείς ότι το προσωπικό είναι ασφαλές όταν παρέχει τη βοήθεια αυτή. Τρίτον, υποδομή ακόμη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρχαν κάποιοι δρόμοι, επειδή δεν έχει γίνει καλή συντήρηση, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε πολύ απόκεντρε, απομονωμένες περιοχές και απαντώ στη δική σας την ερώτηση, ο χρόνος που χρειάζεται για να ταξιδέψει κανείς, για να έχει πρόσβαση σε αυτούς τους ανθρώπους, αυξάνει το περίπλοκο της κατάστασης. Το να υπάρχουν πολλοί εκτοπιστέντες σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει την πρόσβαση στη γη τους, έχουν χάσει την πρόσβαση στην ε, ε, φύτευση. Συνεπώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναρχίσουν από την αρχή και επειδή το είδα εγώ αυτό με τα μάτια μου, οι εταίροι που βρίσκονται εκεί ε, και χρηματοδοτούνται από εμάς κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ορθοποδήσουν και πάλι και να ε, χρησιμοποιήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια το συντομότερο δυνατόν. Παράδειγμα, τι χρηματοδοτούμε εμείς προσπαθούμε ομάδες εκτοπιστέντων ανθρώπων ε, να συγκεντρώνονται σε κάποιο είδους συνεταιρισμού, να τους δίνουμε μία ένα κομμάτι γης το οποίο είναι κοινό και να τους δώσουμε τους σπόρους και κάποια πολύ βασικά εργαλεία για να μπορέσουν να φυτέψουν, για να μπορέσουν να, έχουν, ε, να κάνουν τη συγκομιδή μετά και να μπορέσουν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους χωρίς να χρειάζονται υποχρεωτικά ανθρωπιστική βοήθεια τέτοιου είδους ε, ε, projects ε, έχουν και ένα ακόμη πλέον έκτημα γιατί υπάρχουν συχνά εκτοπιθέντες που, εκτοπιθέντες οι οποίοι προ, προέρχονται από διαφορετικές ε, ε, εθνότητες όπου υπάρχει μια ε, συνεπώς ευκαιρία οι άνθρωποι αυτοί να συνεπάρξουν ειρηνικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν πόσο χαρούμενοι ήταν που υπήρξε μια ελπίδα να μπορέσουν να ξαναρχίσουν κάπως τη ζωή τους, τη δουλειά, την ζωή τους κάπου αλλού με ένα μικρό αγροτεμάχιο σε μια διαφορετική κοινότητα. Να ξαναρχίσουν λοιπόν τη ζωή τους από την αρχή. Όπως είπα και στην αρχή, Το Κονγκό δεν είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα συνδυασμό πολλών προβλημάτων που συνδυάζονται και οδηγούν σε μια ανθρωπιστική κρίση. Υπήρξε επίσης ε, ένα ερώτημα κατά πόσο το 1,8 ε, τα 1,8 δις που χρειάζονται θα βρεθούν, γνωρίζοντας το πόσες κρίσεις υπάρχουν στον κόσμο που θα μπορούσε κανείς να εύχεται κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το ποσό και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό συνεργαζόμαστε με όλους προκειμένου να υπάρξει ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Αν υπάρξει λοιπόν μικρότερο ποσό από το αναγκαίο, να εξασφαλίσουμε το ότι κάθε ευρώ μετράει και ότι πηγαίνει στους τομείς προτεραιότητας και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το σύστημα του ΟΗΕ να είναι και αυτό παρόν επιτόπου και να μπορεί και εκείνο να κάνει την ιεράρχηση αυτή των προτεραιοτήτων, ποιοι τομείς είναι προτεραιότητα προτεραιότητας που είναι για παράδειγμα η διατροφή και η πρόσβαση στο νερό και ποιοι τομείς, ποιες γεωγραφικές ζώνες ε, ε, αποτελούν ε, ζώνες προτεραιότητας. Τώρα, το ζήτημα της σχέσης με, την ενδεχόμενη, με τον ενδεχόμενο πλούτο της χώρας αυτής, που είναι προφανώς τεράστιος, είναι κάτι το γνωρίζουμε, δεν ανθρωπιστικό ζήτημα. Υπήρξαν βέβαια συζητήσεις κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για τα ανθρωπιστικά ζητήματα να υπάρχει τουλάχιστον μία παράπλευρη εκδήλωση για την υπεύθυνη εξόριξη ώστε να μπορεί ε, ο πλούτος αυτός της χώρας να ε, είναι πιο επωφελής για τους ίδιους του, τους πολίτες. Όμως αυτό δεν είναι ένα ζήτημα ανθρωπιστικό, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να καλυφθεί από άλλους συναδέλφους. Το ζήτημα τώρα της πρόσβασης της ανθρωπιστικής. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα Υπήρξαν κάποια χρήματα αναπτυξιακά τα οποία ήταν διαθέσιμα για τους Κασάι και προσπαθήσαμε να τα ε, διοχετεύσουμε στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη της περιοχής για να μπορέσουμε να ε, δημιουργήσουμε μία υποτυπώδη υποδομή ε, ώστε από ανθρωπιστικής απόψεως όταν κάποιος πηγαίνει σε ένα ιατρικό κέντρο να μπορεί να, υπάρχει, ε, ε, να υπάρχουν νοσοκόμοι, να υπάρχουν κάποια φάρμακα διαθέσιμα. Δηλαδή, προσπαθούμε σε συνδυασμό με τα αναπτυξιακά κονδύλια ε, να συμπληρώνουμε ένα τον άλλον για να έχουμε τον μέγιστο αντίκτυπο. Όσον αφορά τώρα τις εκλογές. Κοιτάξτε. Το μόνο που μπορώ να σας πω σε μια εβδομάδα μίλησα με εκατοντάδε ανθρώπου. αυτό κάνει συνήθως όταν πηγαίνει κανείς σε αποστολή. Ε, ο κόσμος φοβάται εν ώψη των εκλογών ότι μπορεί να υπάρξουν ε, συγκρούσεις. Είναι μια περίοδος αβεβαιότητα για το μέλλον, η προεκλογική περίοδος, οπότε ο κόσμος ε, φοβάται για την ενδεχόμενη αύξηση βία κατά τον επόμενο χρόνο. Για το θέμα τώρα της θεομηνίας ή του κατά πόσο προέρχεται από το ανάνθρωπο αυτή η κατάσταση. Αυτά είναι πολιτικά ζητήματα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εμείς από την ανθρωπιστική πλευρά και βάση των ανθρωπιστικών αργών εμείς δεν μπορούμε να είμαστε να έχουμε πολιτική τοποθέτηση, βλέπουμε τι γίνεται επί αλλά δεν ο ρόλος μας αυτός ε, δεν θα πηγαίναμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι ο δικός μας ρόλος να πει ποιος πρέπει να συλληφθεί και ποιος όχι. Ο κύριος Δέβα διακόπτει, αλλά δυστυχώς εκτός μικροφώνου. Δυστυχώς δεν ακούμε γιατί το μικρόφωνο δεν είναι αναμένο. Δεν είπα αυτό. Να μας πείτε όμως αν ξέρετε ποιος είναι ο υπεύθυνο. Ποιος το, ποιος το άρχισε, ποιος κάνει τι σε ποιον, ποιος ε, πυροβολεί ποιον, ποια ομάδα πυροβολεί ποια ομάδα, δεν είναι δυνατόν να μην το βλέπετε αυτό. Αυτό είναι παράλογο. Απάντηση. Υπάρχουν διεθνείς παρατηρητές στο Κονγκό. Αρκετοί μάλιστα που βλέπουν τι γίνεται. Ξέρουμε τι γίνεται επί τόπου. Όμως δεν θέλουμε να διακυβεύεται η πρόσβαση του κόσμου στην ανθρωπιστική βοήθεια και και στο προσωπικό ανθρωπιστικής βοήθειας που υπό ακραίε συνθήκες παρέχουν τη βοήθεια επιτόπου. Καταρχάς, Υπάρχουν όροι και προποθέσει που μα δεσμεύουν, που μα λένε ότι δεν πρέπει να έχουμε πολιτική τοποθέτηση. Και επίση έχουμε και την ευθύνη ενώπιον των ανθρώπων εκεί να μην ε, ε, ε, διακινδυνεύουμε την έκθεσή τους σε περισσότερη βία. Υπάρχουν άλλοι φορείς, των οποίων αυτό είναι το καθήκον και δεν είναι το δικό μας το καθήκον αυτό. Η περιφερειακή διάσταση τώρα. Το έχω τονίσει αυτό πολλές φορές. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας σε σχέση με την περιφερειακή διάσταση. Μισό εκατομμύριο Κογκολέζοι είναι στις ε, γειτονικές χώρες, θα μπορούσαν μάλιστα να γίνουν και περισσότεροι. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να μην ε, διασώσουμε το Κονγκό γιατί είναι μια τεράστια χώρα και ο αντίκτυπο είναι πολύ μεγάλο και για τι γειτονικέ χώρε. Υπάρχει αντίκτυπο στη Ζάμπια, σε άλλε χώρε. Έχουμε και εκεί παράσχει βοήθεια ε, για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τον αντίκτυπο. Ε, Και βλέπουμε τι γίνεται όταν οι Κογκολέζοι, για παράδειγμα, φτάνουν ε, στην Ουγκάντα ε, και ε, προσπαθούμε αν έχουν χολέρα να αντιμετωπίσουμε τις δραματικές συνέπειες αυτής της ασθένειας. Τώρα, ως προς το ποιος παίρνει τη βοήθεια. Κοιτάξτε, λόγω του πώς λειτουργούμε στην ανθρωπιστική βοήθεια, εμείς συμβαλόμεθα είτε μόνο με υπηρεσίες του ΟΗΕ, είτε με διεθνείς ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι διεθνείς ΜΚΟ μερικές φορές έχουν τοπικούς εταίρους, αλλά δεν περνούν από κυβερνητικές υποδομές. Δεν περνάει από κανένα επίπεδο, ούτε κρατικό, ούτε τοπικό βάση του δικού μας κανονισμού μπορούμε μόνο με αυτές τις δύο μορφές ε, ε, φορέων, ε, στο πλαίσιο του ΟΗΕ δηλαδή και των διεθνών ΜΚΟ, να συνάψουμε συμβάσεις. Και όταν, όταν κάναμε την, όταν αποφασίσαμε τα κριτήρια του, της, της σύμβασης πλαίσιο, αυτό είχαμε αποφασίσει Γι' αυτό ακριβώ υπάρχουν τακτικέ επισκέψει, όχι μόνο από τι κεντρικέ εγκαταστάσει. Υπάρχει ένα γραφείο ε, στη Κινσάσα ε, με κόσμο που είναι επιτόπου συνεχώς και που επιβεβαιώνει συνεχώς ε, ποιο δικαιούχο μιλάει σε ποιον και εξασφαλίζει την υλοποίηση των έργων και το κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι αυτά που πρέπει. Ευχαριστώ. like κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο από την υπηρεσία της Επιτροπής. Ναι. Όχι. Α, πείτε μου ποιος είστε παρακαλώ πριν πάρετε το λόγο. Λέγομαι Μάρκος Νιόρ από την ομάδα για την Κεντρική Αφρική. Δεν έχω κάτι να ρωτήσω. Ο κύριος Ντεβά. Μπορείτε να μας εξηγήσετε σε λίγα λεπτά, σαν εμπειρογνώμονος για το θέμα αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ποιος κάνει τι, τι ακριβώς συμβαίνει και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς δεν είμαι εμπειρογνώμονας για την ε, χώρα αυτή. Έχω συναδέλφους που είναι πιο αρμόδιοι από μένα. Αυτά. Okay, we understand it. Ναι, ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε. Κρίμα που ο αρμόδιος που θα έπρεπε να είναι εδώ λείπει. Εν πάση περιπτώσει, με αυτή την τελευταία παρέμβαση ολοκληρώσαμε και το σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Καπινάρα. the next item, Το επόμενο σημείο είναι το σημείο 16, που είναι η καταπολέμηση των παραποιημένων φαρμάκων. Εδώ έχουμε εμπειρογνώμονες. Έχουμε τον καθηγητή Γκεντιλίνη. ο οποίος ε, είναι υπεύθυνος ε, διευθυντής ε, του Ιδρύματος ΣΥΡΑΚ για την πρόσβαση σε καλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη και φάρμακα και τον Μπερνάρ Λερουά. Σας παρακαλώ, ελάτε και οι δύο εδώ στο βήμα.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 στους εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι βουλευτές. Υπάρχουν πολλές ανισότητες, αλλά νομίζω η πιο τραγική ανισότητα είναι αυτή που αφορά την υγεία. Στις 12 Οκτωβρίου του 2009 ο πρόεδρος ε, Σιράκ με τη στήριξη πολλών Αφρικανών ηγετών ξεκίνησε με την πρωτοβουλία της Κοτονού για να σταματήσει η διακίνηση παραποιημένων φαρμάκων, πλαστών φαρμάκων και προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τους ηγέτες ε, του βιομηχανοποιημένου κόσμου για αυτό το φαινόμενο. Ήταν μια πολιτική έκκληση. Την ίδια ώρα βλέπουμε όμως ότι έχουν παραλύσει οι διεθνείς οργανισμοί, ιδιαίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πριν από 8 χρόνια το Συμβούλιο της Ευρώπης πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει με την σύμβαση Medicrim με σκοπό να ποινικοποιήσει τη διακίνηση των πλαστών φαρμάκων. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή περίπτωση διακίνησης πλαστών προϊόντων που πλήττει την υγεία όλων μας σε όλες τις υπήρους συμπεριλαμβανομένες και της Ευρώπης. Βεβαίως ιδιαίτερα πλήττονται οι πιο φτωχές χώρες, είμαστε όμως όλοι ευάλωτοι μπροστά στη διακίνηση και την εμπορία αυτών των πλαστών φαρμάκων. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα αυτό το έγκλημα, το φαρμακευτικό έγκλημα συνεχίζεται. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα που η Επιτροπή σας μετά από την πρωτοβουλία του Λουί Μισελ και του Ιδρύματος ΣΥΡΑΚ πήρε την απόφαση να ενδιαφερθεί για αυτή τη μάστιγα που πλήττει όλους τους ασθενείς, αλλά ιδιαίτερα τους φτωχότερους ασθενείς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα επίσης που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται με δύναμη κατά αυτού του εγκληματικού εμπορίου. Θα σας δείξω κάποιες εικόνες και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι βεβαίως κάποια από αυτά τα φαινόμενα είναι γνωστά Σήμερα υπάρχουν φάρμακα που πολλούνται στις υπαίθριες αγορές και που οδηγούν σε ακαριό θάνατο. Ξέρετε ότι ο τραγουδιστής Prince είναι θύμα ενός πλαστού φαρμάκου. Αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν έχει γίνει γνωστό ευρέως στο κοινό. Και θέλουμε να συνειδητοποιήσετε όλοι ότι όλες οι κατηγορίες, οι κοινωνικές και όλες οι χώρες μπορεί να πληγούν από αυτά τα πλαστά φάρμακα. Θέλω να σας υπενθυμίσω επίσης ότι στον κόσμο πιστεύουμε, και βεβαίως αυτό είναι μια εκτίμηση, περίπου 700 με 800 χιλιάδες νεκροί. Πιο πολύ από τους νεκρούς εξαιτίας ελαιονοσίας. Και αυτό οφείλεται σε πλαστά προϊόντα, ιδιαίτερα σε περιοχές που πολλούνται στην Αφρική, 30 με 70% αυτών των φαρμάκων πουλούνται στην Αφρική και πολλές φορές μέσω του διαδικτύου. Πιστεύουμε ότι αυτό το εμπόριο, αυτή η διακίνηση αποφέρει πολύ περισσότερα από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών Βεβαίως ε, αυτά τα πλασταφάρμακα παράγονται στην Ασία κυρίως, στην Κίνα, περνούν μέσω της ε, Λατινικής Αμερικής και βεβαίως επανέρχονται στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη και στην Αφρική. Η Αφρική όμως δεν είναι όπως ήταν παλιότερα ο κύριος στόχος αυτού του εμπορίου. Σήμερα βλέπετε, κοιτάξτε αυτή τη διαφάνεια, ότι και η Ευρώπη πλήττεται από αυτό το παράνομο εμπόριο. Θέλω να σας υπενθυμίσω ποια είναι η δράση των διεθνών οργανισμών. Ποια είναι η αδυναμία αυτών των διεθνών οργανισμών και η απραξία τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, νομίζω το 1988, συνειδητοποίησε το φαινόμενο στη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στη Γενέβη. 18 χρόνια όμως απόλυτη σιωπής, ένοχη σιωπής ακολούθησαν. Κατόπιν, στη Βηρητό, με την έκκληση των ε, αρχών υπευθύνων για τον τομέα της υγείας, η γαλλόφωνοι υπεύθυνοι στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας ξεκίνησαν τότε με την έκκληση της βιριτού. Ο Ζακ Σιράκ είπε ότι πραγματικά η υγεία είναι ένα καθοριστικό αγαθό και είναι το καθοριστικό στοιχείο για την ανάπτυξη. Βλέπετε με μαύρο χρώμα την περίοδο σιωπής και απραξίας των διεθνών οργανισμών. Σιγά σιγά έχει ξεκινήσει μια συνειδητοποίηση του φαινομένου αυτού. Η Ευρώπη έχει αναλάβει ευτυχώς μια δράση και το 1900, 2011 έχουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά το θέμα αυτό και ακριβώς πριν υπεγράφει στη Μόσχα η σύμβαση Medicrim. Πρόκειται για μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία βεβαίως είναι ανοιχτή για όλες τις χώρες. Ξέρουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός χωρών έχουν υπογράψει. Δυστυχώς όχι αρκετάς, αρκετές χώρες και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν έχει υπογράψει ακόμα, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει και άλλες χώρες στο να υπογράψουν τη σύμβαση αυτή. Παρουσίασα μία έκθεση πριν από λίγα χρόνια, μία έκθεση η οποία έχει υπογραφεί από τις τρεις ακαδημίες στη Γαλλία, την ιατρική, φαρμακευτική και ιατρική, γιατί όπως ξέρετε η παραποίηση των φαρμάκων αφορά επίσης και τα κτηνιατρικά φάρμακα και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Αφρική γιατί 60% των κτηνιατρικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην Αφρική είναι πλαστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αρχές ε, της φαρμακευτικής ιατρικής και της κτηνιατρικής στη Γαλλία, οι τρεις ακαδημίες, αλλά και διεθνείς ακαδημίες, ενδιαφέρονται σήμερα για το θέμα αυτό και στηρίζουν τη δράση μας. Ο κύριος Λερουά πιστεύω ότι θα επανέλθει στο θέμα του Medicrim, της σύμβασης αυτής, η οποία, επαναλαμβάνω, υπεγράφει στην ε, Μόσχα το 2011 και είναι το πρώτο νομικό εργαλείο που ποινικοποιεί τη διακίνηση και τους διακινητές και λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη θυμάτων. Υπάρχουν 11 κυρώσεις από μέρους των κοινοβουλίων και την 1η Ιανουαρίου του 2016 έχει υπογράψει και η Κουινέα και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η σύμβαση αυτή. Είναι πολύ σημαντικό για τις φτωχότερες χώρες και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η διακίνηση αυτών των φαρμάκων θα πρέπει να σταματήσει με τον έλεγχο των σημείων πώλησης και με την μείωση των τιμών των φαρμάκων, χωρίς βεβαίως να αλλοιωθεί και να μειωθεί η ποιότητά τους. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει υλοποίηση της υπόσχεσης για την καθολική ιατρική περίθαλψη, κάτι που δυστυχώς δεν ισχύει σε όλες τις χώρες. Στη διαφάνεια βλέπετε τον ε, Γάλλο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχα την τιμή να παρουσιάσω το θέμα αυτό για 10 λεπτά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τι ήθελα να τον ευαισθητοποιήσω όσον αφορά τα πλαστά φάρμακα, τα παραποιημένα φάρμακα και να τον ρωτήσω αν μπορεί να ενσωματώσει το θέμα αυτό και να το αναφέρει στην επόμενη επίσκεψή του στην Ουαγκαντούγκου. Το έκανε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό που ένας πολιτικός ηγέτης έχει πάρει θέση. Αυτό θα πρέπει βεβαίως να επαναληφθεί, διότι το δράμα των πλαστών φαρμάκων που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και όπως σας είπα και στην αρχή της παρουσίασής μου, επιθυμώ να συνεισφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο επόμενος είναι ο κύριος Λεγουά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να παίρνω το λόγο σήμερα στην Επιτροπή σας. Είμαι διευθυντή του ΙΡΑΤΜ που είναι το ερευνητικό, ε, το ερευνητικό Ινστιτούτο για την ε, παραποίηση των φαρμάτων. Προσπαθεί να έχει μια σφαιρική θεώρηση του προβλήματος ε, για να βελτιωθούν οι νομοθεσίες, ειδικότερα στην Αφρική και στην Νοτιοανατολική Ασία. Επίσης έχουμε αναλάβει μια δράση εκπαίδευσης από κοινού με τον Διεθνή Οργανισμό Τελωνίων ε, για να ε, μπορούμε να εντοπίσουμε καλύτερα τα φάρμακα αυτά και στις τέσσερις εκστρατείες που έχουμε κάνει με τον Οργανισμό Τελωνίων έχουμε καταφέρει 850 εκατομμύρια ε, παραποιημένα φάρμακα να εντοπίσουμε στην Αφρική. Επίσης έχουμε και προληπτικές δράσεις και δράσεις επικοινωνίας. Το πρώτο μας πρόβλημα, περνάμε στην επόμενη διαφάνεια, είναι το γεγονός ότι υπάρχει συχνά μία σύγχυση και μία νομική θεώρηση του προβλήματος που δεν είναι πάντοτε η σωστή. Ε, εμείς γι' αυτό το λόγο αρχίσαμε να υπάρχουμε, ε, εστιάζουμε περισσότερο στην παραποίηση, όμως στην ε, παραποίηση και τα πλαστά φάρμακα. Δηλαδή, πολλέ φορέ ε, υπάρχει 1% ενεργού συστατικού αντί για 100% και επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αυτή την πραγματικότητα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ε, στην Γενική Συνέλευσή του αποφάσισε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στα πλαστά φάρμακα και όχι τόσο στην παραποίηση, γιατί τα πλαστά φάρμακα αντιβαίνουν επίσης στην πνευματική ιδιοκτησία Εκτός από αυτό υπάρχει και μια κατηγορία στην οποία έχουμε περισσότερα προβλήματα. Είναι τα μη αδειοδοτημένα φάρμακα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια φάρμακα που μπαίνουν κάπου όπου δεν υπάρχει άδεια στην, ε, το, για να τοποθετηθούν στην αγορά ε, μέσω παράκαμψης των ε, τελωνίων για παράδειγμα, ένα εμβόλιο το οποίο πρέπει να ταξιδέψει σε 5 βαθμούς θερμοκρασία, όμως ε, ε, βρίσκεται τελικά σε, ένα, ε, σε μια αποβάθρα της Αφρικής σε 60 βαθμούς και συνεπώς ε, δεν, τα στελέχη που υπάρχουν μέσα δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν ενεργά και στην τελευταία εκστρατεία που κάναμε εμείς για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Τελωνίου τα φάρμακα αυτά έρχονταν κυρίως από την Ινδία και ήταν τέτοιου είδους φάρμακα, φάρμακα δηλαδή τα οποία δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές των φαρμάκων λόγω, για παράδειγμα, της θερμοκρασίας που ανέφερα προηγουμένως. Μεθ' επόμενη διαφάνεια. Αυτό το σημείο είναι σημαντικό γιατί τα πλαστά φάρμακα προκαλούν το θάνατο, όμως δημιουργεί και ε, ανθεκτικότητα. Ε, για παράδειγμα, αν υπάρξει μία μόλυνση και την αντιμετωπίζουμε με αντιβιωτικά τα οποία δεν ανταποκρίνονται, τα μικρόβια και τα βακτήρια ενισχύονται λόγω αυτή τη διαδικασία και συνεπώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε δημιουργήσει μικροβιολογική αντοχή. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, επειδή γίνεται κατάχρηση συχνά των αντιβιωτικών, όμω τα πλαστά φάρμακα ενισχύουν αυτό το φαινόμενο. Το είπε και ο κύριος, ε, ο καθηγητής Τιλίνη είπε ότι είναι μια πολύ επικερδής ε, ε, επιχείρηση αυτή, είναι πάρα πολύ ελάχιστες οι κυρώσεις, 6 με 60 ημέρες φυλάκισης στην Αφρική. γιατί δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με το θέμα της δημόσιας υγείας που είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη στην καταστολή αυτού του λαθρεμπόριου πλαστών φαρμάκων. Είναι το βασικό καρτέλ του ε, Μεξικού, το Σιναλόα, όλο και περισσότερο ε, κάνει τη μετάβαση από τα ναρκωτικά στα πλαστά φάρμακα. Όμως, υπάρχει ε, μία πλέον τοξικομανία φαρμάκων, ε, είτε περνάει κανείς από ένα ροζ σε ένα μπλε φάρμακο στην ε, ε, Σαουδική Αραβία, γιατί μπορεί να αποκεφαλιστεί αν πάρετε για παράδειγμα κοκαίνη στην Σαουδική Αραβία, όμως αν πάρετε ένα ροζ ή ένα μπλε χαπάκι δεν θα σας συμβεί, σας τίποτε. Ε, κάτι το οποίο βέβαια ε, έχει ως αποτέλεσμα να, ενισχύονται και οι συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων που γνωρίζουμε πάρα πολύ καιρό. Ε, είναι όλα αυτά λοιπόν πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι. Η κίνδυνη είναι πολύ μεγάλη. Οι δικαστές δεν γνωρίζουν αυτό το θέμα. Συχνά αντιμετωπίζουν ε, υποθέσεις ε, με έναν τρόπο έτσι αρκετά συνηθισμένο και έτσι είναι σε δύσκολη θέση όταν πρέπει να επιληφθούν μια τέτοια υπόθεση. Εγώ είμαι δικαστή σε μια προηγούμενη ζωή και ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργούν. Όμως το λαθρεμπόριο αυτό είναι διακρατικό. Ε, υπάρχουν επιτροπές πλέον διεθνείς που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Είναι δύσκολο όμως. Πήγα ε, στο Πεκίνο, είδα το Γενικό Εισαγγελέα της ε, Κίνας που μου είπε ότι ποτέ δεν ήρθε σε επαφή μαζί του κανείς ε, από την Αφρική. Όμως στην Αφρική υπάρχει πληθώρα αυτών των πλαστών φαρμάκων που προέρχονται από την Κίνα. Πρόκειται λοιπόν για ένα μεγάλο πρόβλημα η διαφθορά. Ξέρω έναν ηγέτη της Δυτικής Αφρικής που εξελέγει και πάλι λόγω ε, των χρημάτων που συνέλεξε μέσω αυτού του λαθρεμπόριου πλαστών φαρμάκων που γίνεται στη χώρα του. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα αυτά δίνει μία ε, δυνατότητα ε, ε, μεγαλύτερου φόρτου για, την, ε, για το δημόσιο τομέα, όμως υπάρχει και μία απειλή κατά του κράτους δικαίου, τόσο πολύ το οργανωμένο έγκλημα ε, έχει ενισχυθεί. Υπάρχει το λαθρεμπόριο, ε, μέσω εμπορευματοκιβωτίων, υπάρχει μέσω ίντερνετ ε, το λαθρεμπόριο, υπάρχει... Ε, η αλλαγή της ημερομηνίας εκμετάλλευσης ε, ε, δηλαδή αλλάζουμε την ημερομηνία λήξης και στέλνουμε ένα φάρμακο στην Αφρική. Για παράδειγμα στο, Περού αυτό γίνεται με το χάπι της επόμενης ημέρας ή αντι... αντισυλληπτικά χάπια που έχουν λήξει. Υπάρχει και μία τέταρτη πρακτική ε, και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να σας το αναφέρω να σας την αναφέρω, να σας επιστήσω την προσοχή σε αυτό το γεγονός. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων. Τα ευρωπαϊκά όργανα δημιούργησαν μια οδηγία ε, πάρα πολύ καλή, ε, βέβαια, η οποία τυποποιεί τις προσεγγίσεις στην Ευρώπη και καλύπτει όλες τις πτυχές. Σε αυτές τις διατάξεις δημιουργούνται Περισσότερε δυνατότητε όσον αφορά τι παράλληλε εισαγωγέ. Τι θα πει αυτό. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα χρήση άλλων διανομέων και των διανομέων από του διανομή του διαπιστευμένους των εργαστηρίων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι τιμέ παραμένουν υψηλέ. Όμω η Ιταλική μαφία και η Ναπολιτάνικη ε, μαφία είδε ε, το κέρδο που θα μπορούσε να έχει από αυτό. Κλέβει 38 τόνων φορτηγά πραγματικών φαρμάκων και τις μεταφέρει σε μερικές χώρες ε, ε, ανατολικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί διανομής ε, ψεύτικη διανομής ανακυκλώνουν αυτά τα φάρμακα για να εξασφαλίσουν τη διανομή τους ε, στις χώρες της δύση σε βάση αυτής της ευρωπαϊκής οδηγίας. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, ότι γίνεται μια αναδιαμόρφωση των φαρμάκων. Μου λέτε, μα είναι πραγματικά φάρμακα τα οποία έχουν κλαπεί. Ναι, εντάξει. Όταν είναι όμως υγρά ε, με ένα λίτρο, κάνουν φάρμακα 100 λίτρων. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, Υπήρξαν τέτοιου είδους πλαστά φαρμακεία, ε, συγγνώμη, φάρμακα στα φαρμακεία, στα πραγματικά φαρμακεία ένα φαρμακείο κατά του καρκίου, το ΙΣΕΠΤΑ, το βρήκαμε ε, εντελώ ε, διαλυμένο, παραποιημένο σε ένα πραγματικό φαρμακείο της Γερμανίας. Πηγαίνετε στο site μας, εμείς κάνουμε μία ανακοινωθέν τύπου ε, στο iratme.com κάθε εβδομάδα, θα δείτε τι δείχνουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις και στη Φιλανδία και στη Δανία Πρέπει λοιπόν ε, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι λιγότερο ιδεαλιστικά ως προς αυτά τα θέματα και να ανησυχήσουν με αυτές τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να αφορούν σύντομα όλες τις χώρες της Ευρώπης. Συνεχίζω. Επόμενη διαφάνεια για ποιο λόγο η καταπολέμηση είναι τόσο λίγο αποτελεσματική. Γιατί οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται. Εμείς ε, κάναμε ένα τουρ ε, στις χώρες του Μεκόν. Κανένας δεν ήρθε να μας δει, κανένας δεν ήρθε να μας μιλήσει για να έχουμε μια περιφερειακή προσέγγιση του προβλήματος. Έχουν πολλά πράγματα να κάνουν και για αυτούς δεν είναι μια προτεραιότητα. Συχνά δεν έχουν και μηχανισμούς επιτόπου. Οι νομοθεσίες επικεντρώνονται κυρίως στην πνευματική ιδιοκτησία και δεν λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα των καταστάσεων και τον αντίκτυπο το σημαντικό στην υγεία. Ε, σας είπα ότι οι ποινές 6 με 60 ημέρες ε, ή ένα απλό πρόστιμο σε μερικές χώρες είναι γελίες αυτές οι ποινές. Οι δικαστές δεν γνωρίζουν τον τομέα και δεν το διακινδυνεύουν. Είναι μια διακρατική εγκληματικότητα η οποία σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μια πραγματική διασυνοριακή συνεργασία. Δεν καταφέρνουμε όμως να την ε, έχουμε αυτή τη συνεργασία. Συνοψίζοντας, δεν επαρκεί να ασχολούμαστε μόνο με την παρατήρηση ή τα πλαστικά... Τα φάρμακα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε γιατί έχει σοβαρές συνέπειες ε, στην δημόσια υγεία. Η εθνική νομοθεσία πρέπει να είναι πλήρης και αποτελεσματική επί τη ε, το, τη σύμβαση με την ΚΡΙΜ ε, γιατί, γιατί αναφέρει τι είναι αυτό που πρέπει να συμπεριλαμβάνει νομοθεσία. Πρέπει να υπάρχει σαφής ορισμός, προσαρμοσμένος, να υπάρξει μια εναρμόνιση των λεπτομαριών ε, των φαρμάκων, μια εναρμόνιση των ποινών, ενίσχυση των ερευνών και διασυνοριακή συνεργασία οι δικαστές είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να εκπαίδευθούν και να τους δοθούν κίνητρα. Εγώ ασχολήθηκα με τα ναρκωτικά 40 χρόνια το 70 ε, δεν είχαμε να κάνουμε και πολλά. Ε, στην αρχή τουλάχιστον μπορούσαμε απλώς να βρούμε το χρήστη των ναρκωτικών. Μετά μπορούσαμε να βρούμε, στο, στο τέλος ε, όταν εξελίχθηκε η όλη διαδικασία, μπορούσαμε να βρούμε και από πού είχαν έρθει τα ναρκωτικά, να φτάσουμε μέχρι τους λογαριασμούς αυτών των ανθρώπων. Την ίδια διαδικασία μπορούμε να ακολουθήσουμε. Και για τα φάρμακα διακυβόβονται τεράστια ποσά είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τις διεθνείς πτυχές και πρέπει να ασχοληθούμε και με τα χρήματα τα οποία αφορά αυτή η διαδικασία γιατί οι χώρες αυτές θα μπορούσαν, οι χώρες πιο φτωχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο και να το καταπολεμήσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντική ε, η, σύνδεση με τις διεθνείς συμβάσεις, ειδικά η MediCream 8 ε, χρόνια έχουν περάσει από την υπογραφή της και ακόμα 20 χρόνια, 20 χώρες μόνο την έχουν ε, κυρώσει. Πρέπει λοιπόν, λοιπόν ακυρωθεί ε, από το μέγιστο αριθμό χωρών και εκτός Ευρώπης. Υπάρχει μία ακόμη σύμβαση του ΟΗΕ, η UNTA, ε, η σύμβαση του Παλέρμο που πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί γιατί αυτή η σύμβαση η οποία υπεγράφει στο Παλέρμο το 2000 είναι ένα σημαντικό εργαλείο, δίνει τα μέσα οργάνωσης μιας πραγματικής διακρατικής συνεργασίας και κυρώθηκε από 180 στα 194 κράτη παγκοσμίω και δίνει τη δυνατότητα διμερούς αντιμετώπισης και δικαστικής συνεργασίας των χωρών. Δίνει τη δυνατότητα λοιπόν συνεργασίας, δίνει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, κάτι το οποίο σημαίνει ότι σε αντίθεση με αυτό που έχει γίνει για αιώνες, ε, ένα ε, ε, κράτος από το οποίο ζητούμε κάποιες πληροφορίες δεν μπορεί να το αρνηθεί και αν το αρνηθεί πρέπει να το αρνηθεί γραπτός και να το αιτιολογήσει. Αυτό βέβαια μας ε, καθιστά, καθιστά μια αλλαγή σε σχέση με άλλους αιώνες όπου μπορούσε να γίνει μια απλή άρνηση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, δίνει τη δυνατότητα ευρύτερη συνεργασίας, δίνει τη δυνατότητα να πάρει κανείς ένα μάρτυρα από μια άλλη χώρα για να καταλάβει καταθέσει σε ένα δικαστήριο μέσα άλλη χώρα Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε μια υπόθεση όπου τρία άτομα εμπλέκονται σε μια σχέση τύπου έγκλημα, ε, οργανωμένο έγκλημα σε πολλές χώρες ε, για μία παράβαση η οποία θα τιμωρηθεί με τουλάχιστον τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Για λιγότερο δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το, τη Σύμβαση του Παλέρμου. Οπότε πρέπει να εναρμονίσουμε λοιπόν την κλίμακα των ποινών και να φτάσουμε σε ποινές που να είναι τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Επόμενη διαφάνεια. Οι κυβερνήσεις μπορούμε να τις μετακινήσουμε ως προς τις απόψεις τους, αλλά πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική, πρέπει να υπάρχει ένας θεσμικός μηχανισμός κατάλληλος, πρέπει να κυρώνουν τις συμβάσεις, πρέπει να εγκρίνουν ε, τις τελευταίες συμβάσεις τις πλέον προσαρμοσμένος και πρέπει να φτάσουν, να πάνε προς τα πίσω και να, να μέχρι να φτάσουν στους υπεύθυνους των εγκλημάτων. Ο το Ινστιτούτο μου έχει προτείνει κάποια υποδείγματα νομοθεσίας που βοήθησαν 7 χώρες αφρικανικές να προσαρμόσουν τις νομοθεσίες τους ε, ένα μενού εστιατορίου δηλαδή ε, σαν να λέμε ένα μενού εστιατορίου που λέει ε, τι νόμοι πρέπει να υπάρχουν για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των πλαστών φραγμάτων. Έχω φέρει USB μαζί μου με πληροφορίες στα γαλλικά, στα αγγλικά ε, και πάρα πολλά άλλα έγγραφα ε, συνοδευτικά. Είμαστε στη διάθεσή σας, αν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας και επί τη βάση όλων αυτών που μπορέσαμε να κάνουμε με κάποιες ε, χώρες της Αφρικής και όσων θα κάνουμε τώρα με τα πέντε κράτη του Μεκόγκ, ελπίζουμε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ομοθεσία και σε άλλα μέρη του κόσμου. Σας ευχαριστώ. <coughs> Okay, thank you. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Ποιος θέλει το λόγο, η κυρία Κέγκε. πολέμηση της ε, απάτης και τις παραποίησης θα πρέπει να είναι στο, στο οποίο δεν καλύπτει δυστυχώς τη δημοσία υγεία. Και για να καταλάβω, για πέστε μου δεν θα έπρεπε να αρχίσει και εξαρτώνται από τέτοια φάρμακα που έρχονται από το εξωτερικό. Αυτό είναι θέμα ανάπτυξης. Εκεί, στις χώρες... Έτερος. Κύριος Βέντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Για πετε μου κάτι όσον αφορά τις φαρμακοβιομηχανίες Τι γίνεται με την εταιρεία που έχει την έδρα της στην Ευρώπη, αλλά το εργοστάσιο στην Ινδία. Να το πρόβλημα. Πρόκειται για τη διαφθορά που έχει διεθνή χαρακτήρα. Έχουμε επίσης και τη διαφοροποιημένη τιμολόγηση. Μια τα όσα μας είπατε θα πρέπει να τα μάθουν όλες οι κοινοβουλικές επιτροπές. δεν είναι μόνο το θέμα της πρόβλησης στα φάρμακα. Είναι το θέμα γενικά των αναπτυσσομένων χωρών. Είναι θέμα και των πόρων που πηγαίνουν στον τομέα της υγείας και στις χώρες εκείνες που βοηθούμε και αυτές πολλές φορές εξάγουν τα φάρμακα που παράγουν σε εμάς. Άρα μπερδεύονται τα πράγματα. Τέλο πάντων, για όλε τι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ μα είναι χρήσιμα αυτά τα οποία μα είπατε. Η υπηρεσία εξωτερική δράση. Μπα και θέλει το λόγο. Μάλιστα. Με όλα όσα συνταγογραφεί ο κύριο Τζεντιλίνη για τη λύση του προβλήματο. Το θέμα είναι όλα αυτά τα φάρμακα που δεν τα χαρακτηρίζονται από αυτή την κατάσταση γεννόσημα, καινούργια, παλιά, ακριβά, φτηνά, είναι θέμα επομένω πνευματική ιδιότητας. Είναι από το συμφέρον μα. Κάτι να γίνει για φυματίωση, για ε, ελονοσία, αγορά των φαρμάκων. Αφ, ποια είναι το γνωμοθεσία μόνο στις πιο προδεσμένες χώρες. να έχουμε φάρμακο υπαγρύπνηση, να προστατεύουμε τους καταγγέλλοντες, να εναρμονίσουμε τα των φαρμακευτικών μητρών, να εναρμονίσουμε τα των φαρμακευτικών μητρών, και είδαμε μέχρι τώρα το τι μπορεί να κάνουν και τρίτες χώρες στο τομέα των φαρμάκων. Επομένω, λοιπόν, θα πρέπει να πηγαίνουν κατευθείαν στο φαρμακευτικό τομέα τα λεφτά τη Ένωση για αυτέ τι χώρε. και κλπ. Και μιλάμε για το ότι τα 50% των φαρμάκων θα πρέπει να κατευθύνονται στην αγορά φαρμάκων για τι λιγότερε χώρε. Και με μεγάλη προσοχή να υποπτεύουμε το αν πιάνουν τόπο τα χρήματα ελέγχους να κάνουμε, εξωτερικούς και εσωτερικούς. Πώ γίνονται οι προμήθειες σε παγκόσμιο επίπεδο και σε συνεργασία με τους αδέλφους ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας, προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με τις χώρες που έχουν φραγκοβιομηχανία και πώ χρησιμοποιούν τα λεφτά από εκεί για να αγοράσουν ρόν που τα παράγουν και οι πιο φτωχέ χώρε να εντοπίσουν τα συστημικά προβλήματα, τη ρίζα του κακού. Να απαντήσετε αν θέλετε. Να απαντήσω, να απαντήσω. Και ο κύριος Λεωρουά να σας απαντήσει. Στην κυρία Κέγγε. Το τέλειο θα ήταν να παράγονται επιτόπου στη χώρα. Τα βάλουμε καλά πάσα απόπειρα που πρόσφατα έγινε προς αυτή την κατεύθυνση κατέληξε σε αποτυχία. Και οι κοινοί γνώμοι οι πάσχοντες, ε, αμφιβάλλουν για την τοπική παραγωγή και θέλουν εισαγόμενα φάρμακα. Μιλάμε για κάποιους ασθενείς οι οποίοι από την Μαυριτανία πάνε στο Ντακάρ και αναζητούν κατασκευαστές ε, διανομής των ε, αυθεντικών φαρμακών. Ε, αλλά άλλοι πάνε στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες, στην Ιταλία. Και εκεί πάνε να αναζητήσουν το φάρμακο που θέλουν. θα ήταν λοιπον εκείνη η τέλεια λύση. Αλλά ακόμα απέχει αυτό. Να μην έχουμε πια την τοπική παραγωγή των πλαστών φαρμάκων. Των πλαστών. Κίνα, Ινδία, στην Ασία έχουμε τεράστια παραγωγή τέτοιων φαρμάκων και σας πενθυμίζω επίσης ότι ό,τι χρησιμοποιεί η φαρμακοβιομηχανία τώρα ως πρώτη ύλη καθώς σε εκείνες τις χώρες που μπορούν να παραγράψουν το, το καλύτερο αλλά ταυτόχρονα μπορούν σε φτηνή τιμή να προωθήσουν τα πλαστά. Πολύ σημαντικό αυτό και πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Δεν θυμάμαι βέβαια τι ρωτήσατε εσείς, αλλά θα σας πω την Πάντως, είπατε το τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνώ μαζί σας. Μπράβο. Όμως, είναι αποκατευτικό το, το αποτέλεσμα, η επίδοση που όπως και ναι, έχετε δίκιο. Και εάν θέλουμε να κάνουμε ένα οικονομικό έλεγχο θα εκπλαγούμε για τα χρήματα που διατίθενται. Δεν απορροφώνται αυτά τα οποία δίνουμε. Και αυτό είναι παράδειγμα. Και η κοινότητα παρέχει χρήματα για του κανόνε που σεβόμαστε, αλλά υπάρχουν χώρε που χρειάζονται τα φάρμακα, αλλά πια δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους. Επομένω, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι έχουμε πετύχει και που έχουμε αποτύχει. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε ό,τι έχουμε κάνει και ο στόχο μα θα είναι να αποσπάσουμε κάποια ουσιαστικά αποτελέσματα. Δεν έχουν τα χρήματα να βρουν τα ποιοτικά φάρμακα. Πού να πάνε να τα βρουν. Δεν υπάρχουν στην Ήπεθρο τα αντίστοιχα φαρμακεία. Πού να τα βρει ο κόσμο και αγοράζουν ό,τι μπορούν να τους δίνουν. και θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Ούτε επίσης να καταδικάσουμε προβλημάτιστα τους μικροεπιχειρηματίες. Δεν φταίει αυτός. Τελικά φταίει ο πολιτής. Αυτός γίνεται μάλλον πολιτής πλαστών, αλλά αυτός δεν, δεν ξέρει να μπορεί να βρει μια εναλλακτική ε, και να μην πηγαίνει στους απαταιώνες. Για τα υπόλοιπα θέματα θα σας πει ο κ. Λερουά. Με της παραγωγής φαρμάκων επιτόπου είναι κάτι που σήμερα δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι με μεγάλη δυσκολία σε ε, πολιτές στο δρόμο που πουλούσαν παραποιημένα και πλαστά φάρμακα. Ο κόσμος φοβάται, φοβάται τα... Η United λοιπόν έχει μια εξαιρετική δράση, θα πρέπει να τη στηρίξουμε. Στην Ευρώπη αυτό που διαπιστώνουμε δεν είναι να παράγονται πλαστά φάρμακα. Στη Μαυριτανία, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν 27 διανομής. 27 διανομής με μια τόσο μικρή χώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσω όλων οι πολυεθνικές πολλές φορές έχουν τη δική τους επαγρύπνηση, το δικό τους έλεγχο, διότι πλήττονται τα συμφέροντά τους με αυτά τα παραποιημένα φάρμακα. Εμείς στο Ινστιτούτο μας θέλουμε να αυξήσουμε την ευαισθησία και στις εταιρείες των οποίων παραποιούνται τα φάρμακα. Ξέρουμε σήμερα ότι όλη η φαρμακοβιομηχανία και είδατε τι έγινε στην Αμερική για την υπατήτηδα γάμα, είναι όμοιρος γιατί με μία θεραπεία η οποία στοιχίζει χίλια δολάρια την ημέρα και διαρκεί τρεις μήνες, 90 μέρες, πώς μπορεί στην Αίγυπτο, παραδείγματο χάρη, που ο αριθμός των ασθενών των φαρμάκων είναι το κύριο πρόβλημα. Πόσο πια μπορεί να ανέβουν οι τιμές των φαρμάκων και πολλές αμερικανικές φαρμακοβιομηχανίες σήμερα έχουν περάσει σε μία ακραία πολιτική όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ. Ξέρουμε ότι τα υποκατάστατα ηρωίνης, όπως το φεντανίλ παραδείγματος χάρη, έχουν καταστροφικές συνέπειες πυρηνικού τύπου θα έλεγα. Εάν πάρετε δηλαδή ε, προϊόντα που περιέχει το φεντανίλ για να δημιουργηθούν και κάποια άλλα παρεμφερή φάρμακα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το φεντανίλ το οποίο πωλείται μέσω διαδικτύου είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προϊόν. Έχουμε που ζυγίζουν κάτω από 20 γραμμάρια. Έτσι λοιπόν μέσω από... Μέσω ταχυδρομείου περνάνε όλες αυτές οι μικρές δόσεις αυτών των φαρμάκων όπως το φεντανίλ. Στη Γαλλία βλέπουμε με ένα πολύ καλό σύστημα, παραδείγματος χάρη, ή για τη λεύκανση των δοντιών, υπάρχει μια διακίνηση παραποιημένων φαρμάκων και πλαστών φαρμάκων. Όμως, δυστυχώς, η βιομηχανία των παραμοιημένων φαρμάκων έχει πλέον επεκταθεί και σε πολύ σοβαρές πολιτείες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, πυρογνώμονέ μας για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις και τις απαντήσεις του. Συμφωνώ με τον κύριο Βέντα ότι και άλλε επιτροπές θα έπρεπε να γνωρίσουν το πρόβλημα να, ε, και για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εμπειρογνώμονες και συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξή μα στο σημείο δένωσης ε, για το πάνελ υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ για την πρόσβαση στα φάρμακα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκρισίας. Κανονικά θα πρέπει να είναι εδώ ένας ε, εκπρόσωπος των ιατρών χωρίς σύνορα. Είναι εδώ. όλα please, you can Yeah, I was giving time for them to sit τον όσων τον Νοέμβριο του 2016 στο Συμβούλιο ΤΡΙΠ τη Παγκόσμια Οργανώσης Εμπορίου είπε η αντιπροσωπεία μας συζητούσαμε τι γίνεται με αυτό το πάνελ για τα φάρμακα και την πρόσβαση και αυτή την προφορική ερώτηση. Και είπε η αντιπροσωπεία της Ένωσης ότι όσα μάθαμε για τη δημόσια υγεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν συμφωνεί με αυτή την αφετηρία και ανεγνωρίστηκε ότι υπάρχουν ζητήματα συστημάτων υγείας λείπουν κάποιοι ε, ειδικοί με δεξιότητες και δεν υπάρχουν επομένως ε, αποθέματα των φαρμάκων, αλλά ποτέ δεν αμφισβητήθηκε. άρα το πρόβλημα θα πρέπει να το εντοπίσουμε σφαιρικά και έτσι να μπορούμε να βοηθήσουμε την προβληματική για την προτασιμότητα ή στα φάρμακα. Οπότε δεν θα έπρεπε να κατηγορεί η Κομισιόν το πάνελ υψηλού επίπεδου για το ότι δεν αντιμετωπίστηκε σφαιρικά το πρόβλημα. Είναι κοινική Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημόσια υγεία. Δεν θα πρέπει επομένως αυτά τα δικαιώματα να είναι ασύμβατα με τα όσα ισχύουν σε επίπεδο πνευματικών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί ότι θα πρέπει η δημόσια υγεία, ότι αυτά τα συμπεράσματα που μας δεσμεύουν, θα έπρεπε να μας δεσμεύουν, αναφέρονται στο σημείο 18, δηλαδή για την αποδέσμευση του, της τιμής από την τελική τιμή. Από την τιμή του πάνω σε επίπεδο έρευνας και υπάρχει το δικαίωμα του κόσμου σε κάποιες λογικές τιμές των φαρμάκων. Αυτά τα είπαμε εκεί στο Συμβούλιο του ΤΡΙΠΣ. Ακριβώς επιλέξει ότι εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση το ότι είναι σύντονες οι συμφωνίες συμπορικές με την... Είναι γεγονό ότι εμεί προσπαθήσαμε στην τελευταίο γύρω διαπραγματεύσεων να δούμε πώ θα θωρακίσουμε περισσότερο τα δικαιώματα. Ε, Όπω α πούμε, τον υπάρχουν επιπλέον πιστοποιητικά ότι θα πρέπει να υπάρχει παράταση για τα αποκλειστικά δικαιώματα. Ε, και αυτά που είπε το 16 ο Συμβούλιο, τι απέγιναν. Πώ είναι δυνατόν να έχουμε αναθεώρηση των όσων ισχύουν σε σχέση με την ε, πνευματική ιδιοκτησία και αυτά που θέλει η Επιτροπή μας, πού είναι η συνέπειά μας όσον αφορά την πολιτική μας, που θέλουμε ότι θέλει να δίνονται και νόσημες αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά για εκατομμύρια σε αυτές τις φτωχές χώρες η πρόσβαση σε γενώσιμα από Κίνα, Ινδία είναι τα μόνα που θελουμε οτι θελει να δινονται και νοσημες αναπτυσσομενες χωρες αλλα για εκατομμυρια σε αυτες τις φτωχες χωρες η προσβαση σε γενωσιμα απο κινα ινδια ειναι τα μόνο που μπορουν να βρουν για να επιβιώσουν Οπότε είναι τελικά κοινό λόγος, δεν υπάρχει πολιτική συνέπεια και ε, γι' αυτό και χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου. Οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώνονται σε σχέση με αυτή την δήλωση της Ένωσης στο τελευταίο Συμβούλιο Τρίψ στον ΠΟΕ τον Οκτώβριο και κατά εκείνη ε, την ε, συνάντηση είχαμε παραγωγούς σε εκατομμύρια μέσω των κοινοτικών συμφωνιών. Η αντιπροσωπή από τη Βραζιλία είπε το ότι είχαν ολόκληρα πλοία, ολόκληρα φορτία που θα πηγαίνανε στην Βραζιλία και τελικά κατεσχέθησαν σε ασπαθίζει όσον αφορά κάποια φάρμακα που έχουν πάρα πολύ αυστηρή βρεσιτεχνία και τελικά ωφελούνται ιδιωτικοί φορείς οι δημόσιες επενδύσεις δεν αποφέρουν ε, πώς θα έχουμε κάποια πουλα από ασθενείς, ε, πώς θα μπορούμε να έχουμε διάφορες πρωτοβουλίες ε, και περισσότερη διαφάνεια για τα νοσοκομεία. Και όπως είπαμε στην αρχή, αυτό το οποίο σήμερα συζητούμε είναι θέμα τα υιοθετήσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να μας εξηγήσει τι θέσεις πήρε, πώς δικαιολογείται η θέση στον ε, ΠΟΕ της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας θα λάβει υπόψη τα θεμητά δημοκρατικά συμφέροντα και με τρόπο θα μπορέσει να διαρθρώσει τη θέση της και τι συμφωνίες γίνονται. Ε, έχει έρθει σε επαφή με κάποιον φορέα κοινωνία των πολιτών για αυτή τη θέση. Ελπίζω να είναι εδώ κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Αλλά πριν από την απάντηση αυτή, είναι εδώ ο Δημήτρη Έινικελ από του Γιατρού Χωρί Σύνορα που θα πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαίνεν. Θα ήθελα για να σας δώσω κάποιες πληροφορίες, θα ήθελα να πω ότι εμείς πήραμε το 1989 ένα βραβείο Νομπέλ σε σχέση με της, ε, όμως ε, πέρσι μπορέσαμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της υπατήτητας γάμα. Ναι, θα μιλάω λίγο πιο σιγά ο Γενικός Γραμματέας Μπαν Κιμούν ε, δημιούργησε ένα υψηλού επίπεδου πάνελ για την πρόσβαση στα φάρμακα και πρότεινε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη ε, συνοχής ε, στην πολιτική μεταξύ των φαρμάκων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τεχνολογία προσπάθησαν να συνεργαστούν για να λύσουν το πρόβλημα. Δεν είναι η πρώτη φορά όμω που ο γενικό γραμματέα έχει ζητήσει ε, την αντιμετώπιση του προβλήματο τη πρόσβαση και των καινοτομιών που χρειάζονται για όλου του ασθενεί, όλε οι ιατρικέ τεχνολογίε, όλου του ασθενεί, φάρμακα, διάγνωση και θεραπείες. Η και του πώ καλύπτεται για τα φαρμακευτικά προϊόντα στι συμφωνίε των κυβερνήσεων ε, και μεταξύ των νέων δεσμεύσεων που έκαναν ε, ε, στο πλαίσιο της, των στόχων αηφόρου ανάπτυξης οι κυβερνήσεις και στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Το πάνελ παρουσιάκων όπως η διάγνωση, η θεραπεία, τα εμβόλια, βελτίωση της πρόσβασης στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στην Ευρώπη και στις χώρες του ΟΣΑ. Όπως επίσης αναγνωρίστηκε η σύνδεση μεταξύ της έλλειψης πρόσβασης των ιατρικών τεχνολογιών και την αντιμετώπιση των επιγουσών αναγκών ε, των τέλων καινοτομίας ε, για ε, την βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα και στην καινοτομία καινοτομία. Ο πρώην γραμματέας, Γενικός Γραμματέας Βάν Κιμούν ενίσχυσε, ε, μάλλον ε, ενθάρρυνε όλες τις χώρες ε, να αναθεωρήσουν αυτές τις συστάσεις για να μπορεί ε, των χωρών αυτών ε, ήταν ε, και χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και διεθνή φόρα όπως το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα, οι συστάσεις που αφορούν τη διαφάνεια και τα νέα μοντέλες και κάποια κράτη τη Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στεγάζουν αυτές τις φαρμακοβιομηχανίες έχουν, δημιουργούν πολλά εμπόδια λόγω των ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ε, στο πλαίσιο του ΟΗΕ να μην υπάρχει μια επιβάση, ήταν, ήταν η βάση της έκθεσης πρωτοβουλίας του 2017 για τη βελτίωση ε, των... της πρόσβασης των φαρμάκων στην Επιτροπή ΕΜΒΗ και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ε, να εκπληρώσει τις ε, υποχρεώσεις της βάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οργάνωσε μία συζήτηση για το πώς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση σε φθηνά φάρμακα για όλους βάσει των συστάσεων του πάνελ του ΟΗΕ για να υπάρξει μία σύνδεση των ευρωπαϊκών και των διεθνών συζητήσεων για το θέμα αυτό. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξη του, έμειναν στην ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων.

άρχισαν να συζητώνται λοιπόν κάποιες συστάσεις και κάποια απορίσματα σε διεθνές και ε, εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, πολλές από τις συστάσεις για την ε, ύπαρξη νέων κανόνων και στρατηγικών για την προώθηση την καινοτομία συμπεριλήφθηκαν. Το τελεστικό του συμβούλιο συζήτησε το θέμα της πρόσβασης ε, στα φάρμακα του τον Ιανουάριο, ώστε να υπάρξει ένας χάρτης πορείας που θα περιγράφει την εργασία που πρέπει να κάνει ο ΠΟΗ για την περίοδο από το 2019 στο 2019 ως ζήτημα για τις αναπτυσσόμενες χώρες όλα τα κράτη-μέλη ε, της... Ε, Ε, ε, της, του ε, ΟΗΕ συμφώνησαν ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση για το πρόβλημα των στόχων αηφόρου ανάπτυξης. Η Πορτογαλία συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη έκθεση και ε, πολλές άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναφερόταν στις τάσεις αυτές, όπως για παράδειγμα η Ολλανδική δήλωση που έλεγε ότι έπρεπε να συμπεριληφθεί. Όμως ε, η μόνιμη επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τις Βρεσιτεχνίες έρχεται σε αντίθεση με τις συστάσεις αυτές, οπότε πρέπει να γίνουν διευρυντικές συζητήσεις για την έκθεση του πάνελ υψηλού επίπεδου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακατανόητη αυτή η συζήτηση γιατί προέρχεται από τη μελέτη που ζήτησε να γίνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση της φαρμακοβιομηχανίας στην Ευρώπη ε, σε σχέση με τα κίνητρα που δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων. Η σχέση δηλαδή μεταξύ ε, και πρέπει να υπάρξει μία σύνδεση με τη διεθνή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραγνωρίζει και υπονομεύει τις προσπάθειες κάποιων κρατών μελών προσπαθούν να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων και να βελτιώσουν τέλεσμα ένα μελλοντικό πρόγραμμα εργασίας που περιλαμβάνει εξαιρέσεις και περιορισμούς στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και ε, της επιρροής που ασκούν οι ευρεσιτεχνίες στην πρόσβαση στα φάρμακα. Ολοκληρώνοντας, ε, η... τα πορίσματα και οι συστάσεις της έκθεσης ε, είναι από τα φάρμακα, τη διάγνωση και στη θεραπεία ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα επόμενα δύο χρόνια θα υπάρξουν νέες ευκαιρίες για την ε, ενσωμάτωση της βελτίωσης της πρόσβασης στα φάρμακα σε διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς διαπραγματεύσεις και το θέμα της ε, ε, οικουμενικής ε, ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν μια πολύ πιο επικοδομητική και φιλόδοξη θέση όσον αφορά την ανάγκη βελτίωσης πρόσβασης στα φάρμακα και στην καινοτονία και πρέπει να γίνει μια νομίξουμε σε καινοτόμες στρατηγικές σε σχέση με τους στόχους ανάπτυξης του 2030. Οπότε... Ε, χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον που δείχνετε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκθεση αυτή. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να ενισχύσετε την κάλυψη των υποχρεώσεων και των συστάσεων που περιλαμβάνει. Όψη το θέμα της ευρεσιτεχνίας και του κόστους ε, ε, της ε, εφαρμογής των κανόνων της ευρεσιτεχνίας στα φάρμακα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay, thank you, Mr. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Η Σεσίλα. Ευχαριστώ. Για όλα αυτά τα οποία είπατε δεν γνωρίζουμε ότι τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πιο δόκιμη προσέγγιση για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια λύση και να δούμε πώς θα καλύψουμε εκείνους που χρειάζεται να καλυφθούν από την προσβασιμότητα στα φάρμακα. Ε, σε επίπεδο χώρα, σε επίπεδο ένωσης, σε επίπεδο τρίτων χωρών, όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνει απομονωμένα. Θα πρέπει να συνδέεται με κάποιο είδους προσπάθεια και δημοκρατισμού χρήστη. Τις όλες αυτές τις χώρες. η κατάσταση εκεί πήγε, πιέζει. Και τελικά το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσει Είναι περίπλοκο. Α, και κάτι άλλο. Ελπίζω να του ληφθεί υπόψη. Θύματα είναι πιο ευάλωτοι, άρρωστοι. Πολλές φορές άνεργοι και εκεί. Άρα είναι αυτοί οι πιο ευάλωτοι, αυτοί πλήσονται περισσότερο και ακόμη περισσότερο ανήλικοι και γυναίκες. Το είδαμε για την Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία. Δεν μπορούσαν οι ασθένειε του AIDS να έχουν τα φάρμακα που χρειάζονται. Δεν έχουν χρήματα, γιατί δεν έχουν δουλειά. Άρα δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ιατρική αγωγή. Αυτό να... δεν έχουν χρήματα, γιατί δεν έχουν δουλειά. Άρα δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ιατρική αγωγή. Αυτό να μπει κορυφαία προτεραιότητα. Η πιο ευάλωτη. Ηλικιωμένη. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος, η Επιτροπή. Παρακαλώ πολύ, δώστε μας και το όνομά σας. Ευχαριστώ πολύ Ήλπιζα ότι θα ήταν μαζί μου και ένας εκπρόσωπος της DigiTrade, αλλά η κυρία Μπιανκόφσκα όταν αρχικά υπευλήθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό που ασχολείται με την πνευματική ιδιοκτησία. Γι' αυτό και νομίζω τελικά δεν είναι εδώ κάποιος από την